Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. για την έναρξη της Συνόδου της Ολομέλειας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το πρωί με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση για το κλίμα στη Νέα Υόρκη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ε, θα γίνει στη Νέα Υόρκη, όπως είπα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον αρμόδιο επίτροπο, τον οποίο θα ήθελα να καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ στην Ολομέλεια. Έχετε το λόγο, κύριε Επιτροπέ, κύριε Μιγέλα Ρίας Κανιέτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα όσο ετοιμαζόμαστε για την τέταρτη Σύνοδο Κορυφή στη Νέα Υόρκη για τη δράση για το κλίμα και του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Ό,τι αφορά τη δράση για το κλίμα, στι 11 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση προ το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη τη διάσκεψη ε, κορυφή με παρουσίαση του, της πολιτικής μας για το κλίμα και τη δέσμευσή μας ε, να επιταχύνουμε τις δεσμεύσει μας. Και μάλιστα ε, θα ε, είναι στο Συμβούλιο και ο πρόεδρος Τούσκ, κάτι που δείχνει πόσο προσιλωμένοι είμαστε σε μια ανάπτυξη συνεκτικής θέσης και πιο φιλόδοξης. Θέλουμε με αποφασιστικότητα, ενότητα και φιλοδοξία να προχωρήσουμε. Και επίσης να δώσουμε προστιθέμενη αξία με μονομένε δράσει των κρατών μελών. Τα ακόλουθα στοιχεία θα χαρακτηρίσουν τη θέση μα. Καταρχήν, έχουμε σημαντική πρόοδο στην προετοιμασία και ολοκλήρωση τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μα για ε, περιβαλλοντική κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Επίση, ε, θέλουμε να υλοποιήσουμε τι εθνικέ ε, συνεισφορέ με συγκεκριμένα μέτρα και αυτέ δράσει. Και τρίτον, προγραμματισμό και επιτήρηση τη πραγματική υλοποίηση και εν ώψη των στόχων ε, και των προθέσεών μα. Τον περασμένο Ιούνιο, πολλοί ηγέτε στήριξαν τι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέτερη απόψη κλίματο μέχρι το 2050, κάτι που προποθέτει ρήξη και έλευθη ε, αλλαγή τη κοινωνία και τη οικονομία μα. Σημαντική πρόκληση. Και μάλιστα από το 1990 ε, αναβαθμίζουμε συνεχώς τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα και συνεχίζουμε μεταξύ του 1990 και του 2017 μειώσαμε κατά 22% της, της, τα αέρια του θερμοκηπίου. Και μάλιστα με την νομοθεσία ε, με και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέχρι το 2030 θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη μείωση ε, διπλάσια από ό,τι στο παρελθόν μεταξύ του 2020 και του 2030 και μάλιστα υιοθετώντα του στόχο του 2050 και με τον μηχανισμό διακυβέρνηση που έχουμε θεσπίσει θα εξασφαλίσουμε επιτάχυση της διαδικασίας και με σταδιακό τρόπο θα κινηθούμε προς μια ουδετερότητα ως προς το κλίμα. Και θεωρούμε ότι με τους στόχους για το 2030 θα μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου κατά 45% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Αυτός είναι ο δεδηλωμένος στόχος στις εθνικές υποσχέσεις συνεισφοράς. Να μειωθούν δηλαδή μέχρι το 2030 τα καψέρια μέχρι ε, γύρω στο 40%. Και μάλιστα η υλοποίηση των στόχων θα έχει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα και θα εξασφαλίσει τη σωστή μας πορεία μέχρι το 2050. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη χρησιμοποιεί τον προπολογισμό της ώστε οι επενδύσεις να ευθυγραμμίζονται και να συμβάλλουν στους κλιματικού μα στόχου. Έχουμε 20% ε, στόχο ε, mainstreaming του κλίματος στον προϋπολογισμό. Περίπου 200 ε, δισεκατομμύρια ε, μέχρι την περίοδο του 2050 για να διευκολύνουμε τη μετάβαση. Και επίσης στη συζήτηση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει 25% του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή 350 εκατομμύρια ευρώ να αφιερωθούν ε, σε κλιματικές δράσεις και τα υπόλοιπα κονδύλια να συμβάλλουν στους, πολιτικούς μας, στους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Θέλουμε μια μετάβαση προς μια ουδέτερη οικονομία από κλιματική άποψη. Αυτό είναι τεράστια επενδυτική πρόκληση που θα πρέπει να αναλάβουμε στο μέλλον. Θέλουμε να επενδύσουμε σε καθαρή ενέργεια, σε καθαρή κινητικότητα. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες πρώτες ύλε, αλλά και θα μας επιτρέψει να απορροφήσουμε τα καυσέρια που δεν μπορούμε να καταργήσουμε. Θέλουμε βέβαια να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, ε, γιατί δεν αρκεί ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συμβάλλει. Και για να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει εξασφαλίσει κίνητρα και προϋποθέσεις για τους επενδυτές ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους όπως είναι το ε, σχέδιο δράσης κλίματος ε, και οι συναφείς νομοθετικές προτάσεις. Θέλουμε φυσικά να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα και στη μείωση του καυσαερίου και στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Επίσης, έχουμε μια στρατηγική προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και διεθνείς προσπάθειες συνεργασίας, στηρίζοντας τις χώρες εταίρους. Και γι' αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζει ε, την τεχνική και αναπτυξιακή συνεργασία της με τις ε, χώρες εταίρους. Και μάλιστα οι εθνικές συνεισφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, στήριξης σημαντικών τομέων όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, η γεωργία και η δασοκομεία, καθώς και η αγροτική ανάπτυξη. Όχι μόνο είμαστε οι πρώτοι δωρητές αναπτυξιακής ανάπτυξης με 74,4 στο 2018, είμαστε και ο μεγαλύτερος δωρητής κλιματικών ε, κονδυλίων για κλιματικές δράσεις. Πάνω από 40% της παγκόσμιας ε, κλιματικής δράσης και οι συνεισφορές μας από το 2013 διπλασιάστηκαν ε, και ξεπερνούν τα 20 δις ετησίως. Επίσης, θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους παγκόσμιους δωρητές και να διευκολύνουμε τις επενδυτικές, τους επενδυτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης θέλουμε δεσμευτικές εμπορικές ε, συμφωνίες που θα προωθούν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις. Και σίγουρα η αλλαγή του κλίματος είναι παγκόσμιο πρόβλημα και προϋποθέτει παγκόσμια ανάληψη ευθύνη. Εμείς ε, διαδραματίζουμε το ρόλο μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά για να υλοποιήσουμε τους πακροπρόθεσμους στόχους μας πρέπει να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας και να τις επιταχύνουμε. Και για όλα αυτά έχουμε ένα ισχυρό μήνυμα που θα πρέπει να μεταβιβάσουμε στη Σύνοδο Κορυφής. Και σίγουρα δεν τελειώνουν εδώ ε, οι εργασίες μας. Όσο και αν έχουμε ενισχύσει τις φιλοδοξίες μας, όση πρόοδο και αν έχουμε επιτελέσει και όσο και αν έχουμε επιταχύνει τις ενέργειές μας, όλα αυτά τα χρόνια περιβαλλοντική και κλιματική δράση ήταν σημαντικά. Αλλά η σύνοδο κορυφή τη Νέα Υόρκη, το μόνο συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξει είναι ότι χρειάζεται περισσότερε δράσει. Και μετά τι ευρωεκλογέ και τι πολιτικέ κατευθυντήρες γραμμέ τη Ursula von der Leyen είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναβαθμίσει και πάλι τις φιλοδοξίε τη με υπεύθυνο τρόπο ε, και με αμύωτη αποφασιστικότητα και πυγμή. Θα υιοθετήσουμε νέες δράσεις ε, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του παρελθόντος και ε, θα τα αναπτύξουμε στο μέλλον. Θέλουμε μια πιο ανταγωνιστική, ε, πιο κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με συνεργασία και καλλιεργώντας την άμυλα με τους εταίρους μας παγκοσμίως. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περνάμε τώρα στο Σύνοδο Κορυφή για του Στόχου Βιώσιμη Ανάπτυξη. Είναι μείζονο πολιτική σημασία και κλείνει τον πρώτο τετραετή κύκλο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου. Χαιρετίζουμε το γεγονό ότι η αρχική κρατών και κυβερνήσεων με όλου του άμεσα ενδιαφερόμενου για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την πρόοδο τη εφαρμογής του θεματολογίου του 2030 και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να δοθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και πολιτική ηγεσία για να προωθηθεί το θεματολόγιο. Επίσης, θα έχουμε μια πολιτική διακήρυξη με σαφή έκκληση για επιτάχυση των προσπαθειών. Και μάλιστα η διακήρυξη αυτή θα περιλαμβάνει τη δέσμευση της διαφύλαξης ακεραιότητας του θεματολογίου του 2030, υιοθετώντα τους στόχους του 2020. Επίσης, κλιματικές δράσεις με βάση τη συνέργεια του θεματολογίου του 2030 με τη Συμφωνία των Παρισίων. Επίση θα πρέπει να έχουμε πιο ρητή μνήμα περιβαλλοντική προστασία που θα περιλαμβάνει και τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη βιώσιμη παραγωγή ε, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ των βασικών μηνυμάτων ε, της, ε, των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να επιταχύνουμε την παρούσα πρόοδο που δεν αρκεί για να υλοποιήσουμε τους στόχους βιώσιμη ανάπτυξη. Μερικέ φορέ η πρόοδο είναι αρνητική. Αυξάνονται οι ανισότητε, η υπερθέρμανση του πλανήτη, χάνουμε βιοπικιλότητα από διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θέλουμε συντονισμένη και επιταχυνόμενη δράση για να ελοπίσουμε τους στόχους του θεματολογίου του 2030 και της Συμφωνίας των Παρισίων. Και θα ήθελα εν κατακλείδη να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τη συνεχή και αμέριστη υποστήριξή μας ε, στη κλιματική δράση που έχουμε προτείνει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αφήγημα στο παγκόσμιο προσκήνιο και να εθαρρύνουμε τους παγκοσμίους εταίρους μας να έχουν φιλόδοξες κλιματικές ε, φιλοδοξίες ε, και δράσεις. Αυτό περιμένουν από εμάς οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και κυρίως οι νέοι που κοινοτοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο για ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για το μήνυμα που σκοπεύει να διαβιβάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σημαντική αυτή σύνοδο κορυφής της Νέας Υόρκης. Περνάμε τώρα στις ε, ομιλίες των συναδέλφων. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Μαγκίνες, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Λαμβάνοντα το λόγο, ε, θέλω να πω ότι γνωρίζω ότι ο Γενικό Γραμματέα ε, των Ηνωμένων Εθνών έχει ζητήσει ένα σχέδιο δράση και όχι μια ομιλία. Και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε μία ομιλία με τις δεσμεύσεις μας, τις δεσμεύσεις τις οποίες θα τηρήσουμε. Επίσης, γνωρίζουμε ότι παρότι οι ομιλίες μας είναι πάντοτε καλές, δεν έχουμε πάντοτε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Υπάρχουν μάλιστα τέσσερα σημεία στα οποία οπισθοδρομούμε για την βιώσιμη ανάπτυξη, παραδείγματο χάρη, για το θέμα της εξάλληψης της πείνας σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η ΦΑΟ έχει επισημάνει ε, κάνουμε βήματα προς τα πίσω και 20 εκατομμύρια άτομα δεν έχουν αρκετό το φαγητό. Αυξάνονται οι ανισότητες, άρα και ο στόχος υπαριθμών 10 δεν ε, τηρείται όπως θα έπρεπε και για τη βιοπικιλότητα δεν έχουμε ανταποκριθεί στους στόχους ε, που έχουμε θέσει. Επίσης, για το θέμα της πείνας σε ολόκληρο τον κόσμο, θέλω να επιμείνω γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα γιατί πρέπει να έχουμε συνοχή στις πολιτικές μας και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί από εμά γνωρίζουμε αυτό το οποίο έχει αναφερθεί για την βιώσιμη εντατικοποίηση, αλλά πολλοί από εμά δεν ξέρουμε τι ακριβώ σημαίνει και πώ θα εξελιχθεί. Χρειάζονται λοιπόν ει βάθο συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στι Επιτροπέ για όλα αυτά τα θέματα. Και ελπίζω ότι το νέο Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ε, αρχίσει τώρα τη θητεία του, θα δώσει δυνατότητα σε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των επιτροπών. Όσον αφορά το κλίμα, ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και η νέα γενιά μας οθεί προς τα μπρο, μα οθεί να κάνουμε κάτι παραπάνω. Επίση, πρέπει να θέσουμε πρόκληση και στον εαυτό μα και στου νέου, για να είμαστε έτοιμοι για τι αλλαγέ στα μοντέλα κατανάλωση που πρέπει να προωθήσουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτού του παγκόσμιου στόχου, του οποίου μπορούμε να επιτύχουμε. Θέλω να μιλήσω για τους ωκεανούς και για τις εκτάσεις. Έχουμε πολλούς στόχους και πρέπει την επόμενη εβδομάδα στους συναδέλφους μας στα Ηνωμένα Έθνη να τονίσουμε ότι η πολυμέρεια είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, αυτές οι προκλήσεις είναι πιο σημαντικές τώρα παρά ποτέ και θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους τους συναδέλφους για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή αλλαγή και όπως ε, ε, όλοι οι συμμετέχοντες θα τονίσουν αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Μίρια Μντάλη. Thank you, Chair. Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το κλίμα είναι βασικό στόχο και η Σύνοδο Κορυφή για το Κλίμα έχει κέρια σημασία για να μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτού ε, του στόχου και αυτέ τι προκλήσει. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσει για ένα ε, σχέδιο για το κλίμα που θα είναι αρκετά φιλόδοξο και θα διασφαλίζει ότι η απαραίτητη μετάβαση θα λάβει χώρα και θα δώσει και του απαραίτητου χρηματοοικονομικού πόρου για να καλύψουμε τι οριζόντιε πολιτικέ που απαιτούνται. Όπω ε, έχει η σημερινή κατάσταση, ακόμη και αν τηρούσαμε πλήρως τις δεσμεύσεις μας για το 2030, πάλι δεν θα ήμασταν, ε, θα πληρούσαμε το στόχο για τους στόχους του Παρισιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθήκον να δείξει φιλοδοξία μέχρι το 2030, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το νέο όραμα για ένα περιβάλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα, ένα καθαρό περιβάλλον. Θέλουμε να έχουμε τα κατάλληλα σχέδια δράσης που θα δείχνουν πώς θα επιτύχουμε τις στρατηγικές που θα έχουμε θεσπίσει και πώς θα τις χρηματοδοτήσουμε. Απαιτούνται αλλαγές στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευών, της βιομηχανίας, της γεωργίας, της δασοκομείας. Η αλλαγή του κλίματος είναι μια πρόκληση για ολόκληρο τον πλανήτη και πρέπει οι λύσεις να αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη, όπως είπε και ο ίδιος ο Επίτροπος. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να παίζει τον ηγετικό ρόλο που έχει Παρέχοντα υποστήριξη στις πλέον ευάλωτε χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε συλλογική δράση. Και ως μέλος της ε, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σύνοδο Κορυφή, θέλω να έχουμε μία ισχυρή φωνή διότι αν έχουμε αδύναμες δεσμεύσεις θα υπονομεύσουμε τις ε, ίδιες μας τις περιφέρειες, τα παιδιά μας, τους λαούς μας. Και μόνο με πραγματική ηγετική δράση μπορούμε να επιταχύνουμε τις ενέργειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους για το κλίμα και δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φοβηθεί σε σχέση με τις ευθύνες που έχει αναλάβει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Το λόγο έχει τώρα η Μαρία Σοράγια Ροντρίγκε Ράμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όντως οι κλιματικές αλλαγές ε, φαίνεται ότι δεν είναι θέμα ιδεολογικό, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε άμεσα, κατεπηγόντως, ε, υιοθετώντα δράσει και αποφάσει άνευ προηγουμένω στην ιστορία μα. Αν ε, δεν αναλάβουμε τέτοιε ρηξικέλευτε δράσει, ο κόσμο κατευθύνεται προ μια υπερθέρμανση πάνω των τριών βαθμών Κελσίου προ τα τέλη του αιώνα και θα έχουμε χάσει οποιαδήποτε ευκαιρία για δράση. Τώρα όμω έχουμε ακόμη χρόνο. Γι' αυτό και η έκκληση του Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πιο σημαντική των Ηνωμένων Εθνών, σε μια σύνοδο κορυφή για την κλιματική δράση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σημαντική αυτή η έκκληση του Γενικού Γραμματέα. Η Σύνοδος κορυφή λαμβάνει χώρα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ένα χρόνο μετά που τα συμβαλόμενα μέρη της Συμφωνίας των Παρισίων καλούνται να υποβάλουν συγκεκριμένες δράσεις και δεσμεύσεις για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για να αποτρέψουμε αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας και το 2050 να μην υπερβούμε τον 1,5 βαθμό αύξηση της θερμοκρασίας. Και μάλιστα όλα αυτά γίνονται μια στιγμή και μια χρονιά που γίναμε μάρτυρες ε, των, της ξηρασίας, ε, των πλημμυρών, ε, των πυρκαγιών που είναι απόρριες αυτής της υπερθέμασης. Φυσικά, η Σύνοδος Κορυφής δεν είναι για να ε, εκφωνούνται στον φόδι ομιλίε, αλλά για να προετοιμαστούν συγκεκριμένε δράσει και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευθεί υπέρ μια κλιματικά ουδέτερη δράση ε, εν ώψη του 2050. Και μάλιστα η υποψήφια πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε την πρώτη κλιματική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πολύ φιλόδοξο έργο και προϋποθέτει και κατάλληλο προπολογισμό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μετατραπεί σε κλιματική τράπεζα. Επίσης, ε, ε, μια και θα λάβω μέρος στην ε, Σύνοδο Κορυφή, ω μέλο στην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι στα πλαίσια της πολυμέρειας μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία της αλλαγής και ειλικρινά πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο, σε, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπάς Έκχοτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Επίτροπε, την Παρασκευή θα έχουμε την ε, αρχή μιας εβδομάδας δράσης, ε, παγκόσμιας δράσης. Ε, πάρα πολλοί πολίτες θα κατέβουν στους δρόμους. Νομίζω το έχουμε πει αυτό αρκετές φορές. Αλλά θέλουμε πολλές περισσότερες δράσεις από αυτές που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Επίτροπε, προφανώς αυτή θα είναι μία από τις τελευταίες σας αλλά θα πρέπει να έχετε δει στις σημειώσεις σας ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα στην Ευρώπη ε, όσον αφορά το κλίμα. Ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε την ε, ουδετερότητα όσον αφορά στον άνθρακα, αλλά ακόμα δεν το έχουμε επιτύχει. Πιστεύω ότι αυτή είναι κατ' ουσίαν ομιλία που θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλουν περισσότερη δράση. Οι πολιτικοί να ακούν την επιστήμη και αυτό δεν γίνεται και η επιστήμη είναι απόλυτα σαφή. Έχουμε 10 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι προετοιμαζόμαστε για μια νέα οικονομία και από αυτού πρέπει να είμαστε από αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει υψηλότερε φιλοδοξίε, άρα υπάρχει κάποια αλλαγή, ενδεχομένω και στην Επιτροπή, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώ θα πούν, τι θα κάνουν σχετικά με την νομοθεσία για το κλίμα. Εκεί έχουν σημαντικό ρόλο. Μιλώντα ε, στου ανθρώπου τη γενική σα διεύθυνση, δεν νομίζω ότι φλέγονται. Λένε θα υπάρξει κάποια κλιματική νομοθεσία και μετά θα υπάρξουν πολλέ διαβουλεύσει για το τι θα ακολουθήσει. Εμεί λοιπόν, λοιπόν περιμένουμε η Ευρώπη να έχει υψηλότερες φιλοδοξίες, τουλάχιστον μείον 5 βαθμούς, την επόμενη χρονιά πριν αρχίσει η συνεδρία στο Παρίσι. Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι, την ελάχιστη αλλαγή, αλλιώς οι άνθρωποι στις διαδηλώσεις στον δρόμο ε, θα απογοητευτούν και πάλι, γιατί δεν θα έχει αναλάβει δράση ο κόσμος και κυρίως δεν θα έχει αναλάβει δράση η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριε Ζωντάν Παρδελά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Αντώνιο Γκουτιέρε, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον περασμένο μήνα μα είπε ότι για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή δεν αρκούν οι ωραίοι λόγοι. Χρειαζόμαστε δράση. Κανεί δεν μπορεί να αρνηθεί σήμερα ότι οι διεθνεί οργανισμοί, Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. φέρουν βαρύ ευθύνη για την κλιματική αλλαγή. Αυτοί οι οργανισμοί ε, άφησαν τις βάσεις ε, ε, της αντιμετώπισης της πολιτικής του κλίματος να πάνε χαμένες. Μιλάμε για δράσεις που χάνει της παγκοσμιοποίησης δεν προώθησαν τα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαμε να παράγουμε σε περιοχές κοντά στα σημεία που ζούμε για την οικολογία, για τους οικολόγους σε όλο τον κόσμο βλέπουμε ότι παντού κυριαρχεί η υποκρισία. Αυτό το οποίο προσπαθούν όλοι να εφαρμόσουν είναι η άρση των περιοριστικών ρυθμίσεων και ε, ξέρω ότι οι θεοί κοροϊδεύουν τους ανθρώπους ε, που δεν τους σέβονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Άννα Ζαλεύσκα. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Στην ομιλία του ο κύριος Επίτροπος μίλησε για φιλοδοξία, για αποφασιστικότητα, για πυγμή. Ευτυχώς μίλησε και για ρεαλιστικές δράσεις. Έχω μία ερώτηση. Είμαστε προετοιμασμένοι για μία συζήτηση μετά από μία ρεαλιστική ανάλυση των δράσεων που χρειάζονται, αλλά και των δυνατοτήτων που έχουν οι επιμέρους χώρες, μέλη. Έχουμε προγραμματίσει ε, Ουσιαστικέ και ρεαλιστικέ επενδύσει για το μέλλον. Για να είναι όλα αυτά ρεαλιστικά και πραγματικά έχουμε πραγματικά μέσα χρηματοδότηση και κατάλληλα κονδύλια. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για πάνω από 320 δισεκατομμύρια ευρώ για τι κλιματικέ δράσει. Ένα τεράστιο ποσό. Η Ευρωπαϊκή όμως Επιτροπή δεν εκπώνησε προπολογισμό για το μετασχηματισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το επισήμανε και προτείναμε μικρό κονδύλιο σχετικά, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ρωτώ λοιπόν, τα, φιλόδοξα ε, σχέδιά σας, αν δεν συνδυαστούν με κατάλληλες οικονομικές δράσεις, ε, μήπως κινδυνεύουν να αυξήσουν αντί να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε τις προδιαγραφές μας και να έχουμε μια οικονομία με υψηλές εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πέτρος Κόκαλης. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Ε, την άλλη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μας περιμένει στη Νέα Υόρκη να παρουσιάσουμε πώς θα, θα σταματήσουμε την αύξηση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα στο 2020 και θα τις μηδενίσουμε ως το 2050. Η φωνή της επιστήμης είναι ενωμένη, είναι ξεκάθαρη και σημάνει συναγερμό ένα συναγερμό που έχει κυριαρχήσει την νεολαία της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Η απάντηση λοιπόν στην κλιματική έκτακτη ανάγκη δεν απαιτεί τίποτα λιγότερο από το ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Και έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να ελοπίσουμε μια τακτική και δίκαια μετάβαση εφαρμόζοντας τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης το πολιτικό πρόγραμμα της συμφωνίας του παρισιού που διεκδικούν ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής την εξάλληψη της φτώχειας και της ακραίας ανισότητας. η πολιτική διακήρυξη του συνεδρίου αναφέρει ρητά ότι ξέρουμε τον κόσμο που θέλουμε και έχουμε τον δρόμο να πάμε εκεί. ας το κάνουμε λοιπόν ενσωματώνοντας στους 17 ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο από το νέο πρόγραμμα που ετοιμάζει ο αντιπρόεδρος τίμερμανς από ένα νέο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο και αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν γίνεται καταψηφίζοντας χτες το ψήφισμα καταδίκης κατά της καταστροφής του αμαζονίου. ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ελεονόρα Εύη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτή τη συζήτηση το πραγματικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ότι ε, δυστυχώς ενισχύουμε τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτή είναι μια πλήρης αντίφαση με τους ε, στόχους ε, που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ψηλότερους, στόχου. ψηλότερους στόχους. 350 εκατομμύρια λέμε, αλλά κατ' ουσίαν χρειαζόμαστε στην Ευρώπη πολλά περισσότερα δισεκατομμύρια. 55 δις θα χρειαζόντουσαν κάθε χρόνο, αλλά αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Στην ε, συνάντηση κορυφή της Νέας Υόρκης θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις να σταματήσουμε τα ορυκτά κάψιμα και να τα εγκαταλείψουμε πλήρω μέσω πρόθεσμα. Να βρούμε έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια, γιατί είναι απολύτως παράλογο να αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο τις, ε, τα μέσα, ε, τα προϊόντα που είναι απολύτως απαραίτητα και αυτά που έχουν σχέση με το κλίμα. Δεν χρησιμεύουν μόνο οι δασμοί. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει η σωστή φορολογία, να υπάρχουν ε, διαφανείς στόχοι όσον αφορά στο κλίμα και όλα αυτά να συμβαδίζουν με την ιδέα των ανοιχτών αγορών του ανταγωνισμού για να επιβραβεύουμε πραγματικά εκείνους οι οποίοι κάνουν καινοτομίες. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Τομάς Μπε. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι οι ηγέτες στην συνεργασία και στην ανάπτυξη και ο ρόλος αυτός αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία σε αυτές ε, τις ε, εποχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθοδηγήσει τις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών όπως έγινε και με την θέσπιση των στόχων της χιλιετίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και είμαστε περήφανοι για αυτό το οποίο κάναμε μέχρι τώρα και τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή για όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Χαίρομαι διότι η εκλεγήσα πρόεδρος της Επιτροπής φαίνεται έτοιμη να αναλάβει δράση και όλοι οι νέοι επίτροποι θα πρέπει να συνεισφέρουν στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε όμως μια ευρύτερη δέσμευση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Προσβλέπω λοιπόν στη σύνοδο, της, σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας, όπου θα είμαι συμπρόεδρος της αντιπροσωπείας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανοίξει το δρόμο και να κατευθύνουμε την πολιτική προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια και την, την πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η οποία θα είναι σωστά ισορροπημένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Σούντο Μπούλμαν. Micro, μάικρο. Ανάψτε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Colleagues, uh, President, a week ahead of uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, μία εβδομάδα πριν από τη Σύνοδο Κορυφή στη Νέα Υόρκη, οι στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι που όλοι το συζητάνε. Το συζητούν οι επιχειρηματίε, το συζητούν οι πολιτικοί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τι σημαίνει όμω στα αλήθεια. Είμαστε σύμφωνα με τους στόχους μας στο σωστό χρονοδιάγραμμα. Όχι, δεν είμαστε χρονικά σωστοί. Και καθυστερούμε πολύ συχνά λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Δεν λαμβάνονται αποφασιστικές δράσεις και αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά. Ιδίω στις χώρες με χαμηλό εισόδημα χρειαζόμαστε 530 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορεί να φαίνεται τεράστιο ποσό, αλλά αυτό αντιπροσωπεύει μόνο 0,5% του συνολικού ΑΕΠ του πλανήτη. Άρα λοιπόν, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε αυτά τα χρήματα για να έχουμε σωστή θέρμανση, σωστή ίδρευση, σωστές παροχές υγείας, ε, για να μπορούν τα παιδιά στις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου να δίνονται με τα απαραίτητα ρούχα. Ακόμη και αν βλέπουμε κάποια πρόοδο, δεν αρκούν αυτά τα οποία γίνονται. Καταστρέφονται τα τροπικά δάση χάρη της παραγωγής κρέατος. Βλέπουμε ότι τα ενδύματα παράγονται υπό τις χειρότερες συνθήκες ένδυας. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και πιστεύω ότι το κλειδί για τον αγώνα ε, υπέρ των στόχων της ανάπτυξης είναι ο αγώνας κατά της ανισότητας και της αδικίας. Μόνο αν επενδύσουμε στην κοινωνία μας και μόνο ε, αν οι άνθρωποι πάρουν το πεπρωμένο τους στα χέρια τους, να τους βοηθήσουμε να το κάνουν αυτό με ισχυρές επενδύσεις, με πολυμέρεια και με μια πολιτική για καλύτερη εκπαίδευση. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια ευκαιρία στις επόμενες γενιές. Αυτό περιμένουμε από την επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κατρίν Σαμπό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, την επόμενη εβδομάδα κάποιοι από εμά θα είμαστε στη Σύνοδο Κορυφή των Ηνωμένων Εθνών για τι ε, δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα στο Μονακό οι εμπειρογνώμονες για το κλίμα θα παρουσιάσουν ε, την ε, έκθεσή τους για τους ωκεανούς. Μια έκθεση που ζητήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια που φαίνεται ότι είναι αρκετά ανησυχητική. Οι ωκεανοί πραγματικά καίγονται αγαπητοί συνάδελφοι. Οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα συνεχίζονται και οι βασικές ε, υπηρεσίες των ωκεανών στην ε, ανθρωπότητα, χάρη στη φωτοσύνθεση και στους φυτικούς οργανισμούς, οι ωκεανοί δίνουν το ίμιση του οξυγόνου που, ε, θέλουν, που χρειαζόμαστε στον πλανήτη μας. Είναι ο πνεύμονας οξυγόνου για τον πλανήτη μας. Οι ωκεανοί εξασφαλίζουν τα προστοζήν για 3 δισεκατομμύρια κατοίκους η συχνότητα των κυκλώνων αποτελούν συνέπεια της υπερθέρμανσης των ωκεανών. Η έλλειψη οξυγόνου και η οξύνηση των ωκεανών είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία θα μας αποκαλύψει αυτή η νέα έκθεση. Το 2015 στην COP21 στο Παρίσι ακούστηκε η φωνή των ωκεανών. Είναι ένα θέμα το οποίο επιτέλους κινητοποίησε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη χάρη στη δουλειά του Επιτρόπου Βέλλα. Η Χιλή στην, την επόμενη COP25 την έχει ονομάσει ε, γαλάζια COP. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας το θέμα των ωκεανών γιατί αποτελούν και τμήμα της λύσης. Πρέπει να επαναφέρουμε την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, να αναπτύξουμε την θαλάσσια ενέργεια, να προστατεύσουμε ε, τα ενδιατήματα. Γιατί πρέπει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τον ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και περιμένουμε από τον Αντιπρόεδρο που θα είναι υπεύθυνο αυτή τη νέα πράσινη συμφωνία, να είναι πράσινη και γαλάζια συμφωνία και να λάβουμε υπόψη μα του ωκεανού, αναγνωρίζοντά του ω αγαθό τη ανθρωπότητα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Άιλιν Μακλόιτ. Κύριε Πρόεδρε, την Παρασκευή ε, χιλιάδε νέοι θα, πάνε, θα στη Σκοτία αλλά και αλλού θα υπάρξουν διαδηλώσει γιατί θέλουμε οι πολιτικοί να εφαρμόσουν τα φιλόδοξα σχέδια. Πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε πολιτικές που θα καλύψουν τις ανάγκες του πλανήτη. Ως ε, μέλος ε, της Επιτροπής ε, για την συνάντηση για το κλίμα πρέπει να εκπέμψουμε ισχυρό μήνυμα, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, να αναλάβουμε θαλα... θα... πολύ θαλα... θαραλές ενέργειες για να επιτύχουμε τους στόχους. Αυτό ακριβώς περιμένουν οι άλλοι από εμά και ακριβώς εκεί πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Η δική μου η χώρα, η Σκοτία, ήταν αναγκασμένη να ε, κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ε, εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στην κλιματική αλλαγή και θέλουμε να ε, βοηθήσουν όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν έτσι ώστε να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηθικό καθήκον να καθοδηγεί την όλη διαδικασία, να έχει φιλόδοξους στόχους. Η Σκοτία θα προσφέρει την υποστήριξή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σίλβια Λίμερ για ένα λεπτό. Το Δεκέμβρη είχαμε πάλι αυτό το και θα έχουμε το τσίρκο του κλίματος ε, ε, όπου όλοι αυτοί θα μαζευτούν για να συζητήσουν για το κλίμα ε, αλλά εντωμεταξύ όλοι θα πάνε εκεί διανύοντας πάρα πολλά χιλιόμετρα και θα εκπέμψουν τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Άρα δηλαδή μιλάμε για υποκρισία, απόλυτη υποκρισία. Υποτίθεται θέλουν να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε και την διασπάθηση των εκατομμυρίων ευρώ, τα χρήματα του φορολογουμένου. Ας μην τα αναφέρουμε και αυτό. Ενώ λοιπόν αυτοί που ασχολούνται με το κλίμα πάνε σε ωραίε πόλει, στο Μαρακέ, ε, στο Λίμα, στο Περού, στη Νότια Αφρική, στο Μπαλί το 2007 και πολλέ σε πολλέ άλλε πόλει. Εν τω μεταξύ όμω τι γίνεται, ανακαλύπτουν υποτίθεται κασάνδρε και στι πατρίδε του προσπαθούν να εμποδίσουν του απλού πολίτε ε, να πετάνε με το αεροπλάνο, περιορίζουν τα μέσα μεταφορά ε, και του απαγορεύουν και την χρήση κακού κρέατος. Έτσι τα αναφέρω αυτά ενδεικτικά. Βεβαίω, ε, θέλω να σα πω ότι εγώ θα πάω το Δεκέμβρη στη συνάντηση, αλλά το διοξείδιο του άνθρακα, να σα πω κάτι, δεν είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτά είχα να σα πω για σήμερα και θα επανέλθω. Χαίρετε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Γιατβίγκα Βυσνιεύσκα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σήμερα ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πιο φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική στον κόσμο. Δεν θεωρώ ότι στη Νέα Υόρκη θα πρέπει να κάνουμε και νέες διακηρύξεις για την αναβάθμιση των φιλοδοξιών μας. Γιατί η υπερβολικά περιοριστική περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη προκάλεσε τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει ε, σε, σε πολλούς τομείς ιδιαίτερα στο τομέα του χάλιβα, για παράδειγμα, έχουμε κατακλειστεί από φθηνό κινέζικο χάλιβα. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υπερβολικά περιοριστική περιβαλλοντική πολιτική που οδηγεί σε μετεκατάσταση επιχειρήσεων σε χώρε που έχουν χαμηλότερε προδιαγραφέ. Έτσι αυξάνεται η ανεργία σε εμά και μειώνεται η ανταγωνιστικότητά μα. Οπότε δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και την ενεργειακή ένδυα στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών. 54 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε βρίσκονται στο κατόφλι τη ενεργειακή ένδυα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Εγώ θα ήθελα να προστατεύσουμε το κλίμα, εννοείται, αλλά ο ενεργειακός και κλιματικός μετασχηματισμός θα πρέπει να είναι δίκαιος και να λαμβάνει υπόψη τη, τα διαφορετικά ενεργειακά μείγματα των κρατών μελών. Για παράδειγμα, η Πολωνία έχει ένα ενεργειακό μείγμα με βάση τον άνθρακα. Θέλουμε λοιπόν επαρκή κονδύλια για μια δίκαιη μετάβαση σε θέματα κλίματος και περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σίλβια Μόντιχ για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα ένα προγνώμονας της ένας γνώμονα της ανταγωνιστικότητας ε, είναι η προσαρμοστικότητα. Οι κερδισμένοι ε, θα είναι αυτοί που θα προσαρμοστούν στα όρια των κλιματικών αλλαγών και θα καινοτομήσουν και θα προσαρμόσουν την παραγωγή τους. Μας μιλήσατε κύριε Επίτροπε για μειώσεις ε, αερίων του θερμοκηπίου το 45% μέχρι το 2030 δεν αρκεί. Οι επιστήμονες μιλούν για 55% ανάγκη μείωσης ε, των καυσαερίων. Κάτι που δείχνει ότι οι φιλοδοξίες μας δεν ε, είναι αρκετές. Οι στόχοι μας θα πρέπει να εδράζονται σε επιστημονικά κριτήρια και επιστημονικές συστάσεις και πορίσματα. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανισότητα στα θέματα των κλιματικών αλλαγών και απώλεια βιοπικιλότητας. Ε, δυστυχώς ε, αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς η απώλεια της βιοπικιλότητας. Και η βιοπικιλότητα αφορά την ίδια την ανθεκτικότητα του πλανήτη μας. Ε, ο πλανήτης δεν αντέχει την υπερθέρμανση, δεν αντέχει την αύξηση της θερμοκρασίας. Θα πρέπει λοιπόν, όπως τίποτε, να μειώσουμε τη χρήση φυσικών πόρων, να κάνουμε μεγαλύτερη οικονομία, κάτι που απαιτεί ψηλότερες φιλοδοξίες και καλύτερες δράσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η υποψήφια πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der είπε ότι αισθάνομαι ότι παρασύρομαι από το πάθος και την ενέργεια όλων αυτών των νέων ανθρώπων που διαδηλώνουν στους δρόμους μας. Και θέλω να σας πω ότι υποστηρίζω επιφύλακτα την κυρία Φοντελάιν. Θέλω να ακολουθήσουμε όλοι τον ίδιο δρόμο. Θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι στο κλίμα. Θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 να είναι μάλιστα ακόμα υψηλότερος ο στόχος και να προειδοποιήσουμε ευχαριστήσω όλους ε, ε, να μην προσπαθούν να εξακοντίζουν ύβρις. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση μέχρι τώρα είναι στην αιχμή του δόρατος όσον αφορά την προστασία του κλίματος. Είμαστε μια, ένας μεγάλος οικονομικός ε, σύνδεσμος στην Ευρώπη. Εμείς αποφασίσαμε για εκπομπές στο Παρίσι. Αυτά βέβαια τα έχουμε επιτύχει. Μπορεί να μην φτάνουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Όμως το βλέμμα μας πρέπει να το στρέψουμε σε άλλους που ρηπαίνουν το περιβάλλον και να δούμε πώς θα διεξάγουμε το διάλογο. Πράγματι, να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, αλλά να πηγαίνουμε και πιο πέρα από αυτό. Αυτό δυστυχώ βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει σε πολλέ μεγάλε οικονομίε, άρα πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλή δουλειά. Για να πείσουμε του άλλου, χρειαζόμαστε πολύ δρόμο. Το δρόμο τον έχει καταδείξει η κυρία Φόντερ Λάιν. Τόντι πρέπει να αφαιρέσουμε τον άνθρακα από τη βιομηχανία, να μην αναγκάσουμε τι ε, βιομηχανίε να μετακομίζουν σε άλλε τοποθεσίε. Αν συνδυάσουμε την προστασία του κλίματο και την οικονομία, νομίζω τότε θα μπορέσουμε να είμαστε πρότυπο ολόκληρο τον κόσμο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο ρυθμό των ατόμων που πλήττονται από την ένδυα αυξάνεται συνεχώ. Η απώλεια βιοπικιλότητα είναι ανησυχητική και η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται, απειλώντα και την πολυμέρεια. Ένα χρόνο πριν χρειαστεί να ε, ε, εντείνουμε τους στόχους μας σύμφωνα με τους στόχους του Παρισιού, βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Τα σχέδια τα οποία εφαρμόζονται είναι ανεπαρκή για να αποφύγουν την υπερθέρμανση του κλίματος. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τη στρατηγική μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και για να επαναλάβουμε τις φιλοδοξίες μας για την κλιματική αλλαγή. Η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος ε, είναι σαφή μέτρα και για την καταπολέμηση της ένδυας, της ε, πείνας και είναι πρωταρχική σημασίας τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν να υποστηρίζονται από όλους και να μην επιβαρύνουν μόνο τους πλέον ευάλωτους ε, οικονομικά πολιτισμούς, τόσο στις δικές μας χώρες όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε ισχυρά μέτρα που θα είναι κατάλληλα για να μειώσουν τις ανισότητες και να μην τις οξύνουν. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, χαμηλές φιλοδοξίες. Θα πρέπει να δείξουμε θάρρος και να έχουμε τα μέσα στο μέλλον να είμαστε περισσότερο δραστήριοι. Να μην καθυστερούμε πλέον. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Φρεντερή Κρίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να παραφράσω έναν πρώην Γάλλο πρόεδρο, τον Ζακ Σιράκ, το σπίτι καίγεται. Αλλά σήμερα, 17 χρόνια μετά τη Σύνοδο Κορυφή του Ιωάννεσμπουργκ, η διαφορά είναι ότι ο κόσμο το κοιτάει. Και αυτό θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, χάρη στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρε. Σίγουρα, μα είπε ο Επίτροπο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τηρήσει τι προθεσμίε ε, και του κανόνε τη ε, φιλοδοξία και τη δράση. Και σήμερα έχουμε 23% μείωση των εκπομπών. Κι όμως το 2019 είχαμε επανειλημμένες ε, θεομηνίες, πλημμύρες, ε, καύσονες, πυρκαγιές, ε, κυκλώνες, τυφώνες, δεν αρκεί λοιπόν αυτό που κάνουμε για να τηρήσουμε τη Συμφωνία των Παρισιών. Θα πρέπει να τριπλασιάσουμε τις προσπάθειες, λένε τα Ηνωμένα Έθνη, για να ε, περιορίσουμε την υπερθέρμανση στους δύο βαθμούς και αν θέλουμε στον 1,5 βαθμό θα πρέπει να τις πενταπλασιάσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε τις προσπάθειες και να τις αναβαθμίσουμε. Εμείς στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουμε μόνο το 9% των παγκόσμιων εκπομπών. Θα πρέπει όμως να δείξουμε στους υπόλοιπους, στους βασικούς ε, χώρες, στους βασικούς εταίρους που ρηπαίνουν, στις χώρες που ρηπαίνουν, θα πρέπει να δείξουμε ότι η κλιματική δράση ενισχύει τις οικονομίες και δεν τις ε, ε, και δεν τις υποβαθμίζει και θα πρέπει το οικολογικό σύμφωνο, το Green Deal της ε, κυρίας Φοντερ να γίνει πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Καρίμα Ντελή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο πλανήτης μας στέλνει σήματα εκτάκτου ανάγκης. Καίγεται ο, ο Αμαζόνιος, πνίγεται ο πλανήτης μας. Και όλοι οι επιστήμονες συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα προειδοποιητικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν χρειάζονται πια λόγοι και κενά λόγια. Πρέπει πλέον να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα δράσης. Πρέπει η Ευρώπη να δείξει υποδειγματική συμπεριφορά. Και υπενθυμίζω ότι κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τηρεί τη Συμφωνία του Παρισιού. Ξυπνήστε λοιπόν όλοι. Όλοι οι τομείς θα πρέπει να συνεισφέρουν και πρέπει από τώρα, ήδη από αυτή την εβδομάδα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, να πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ της φορολόγησης των αεροπορικών μεταφορών. Η Ευρώπη είναι σε θέση να το κάνει. Ελπίζω ότι θα επωφεληθείτε της ευκαιρίας, γιατί σας το λέω, αν δεν κάνετε τίποτα, αύριο δεν θα είστε μόνο υπόλογοι, θα είστε ένοχοι αυτής της εγκληματικής δράσης. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα. Το λόγο έχει ο κύριος Πουσαντεύ Γιάλμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι κινδυνολόγοι των κλιματικών αλλαγών επίση ρηπαίνουν περισσότερο από ότι εμά που μας κατηγορούν για σκεπτικιστέ ω προς το κλίμα. αυτό το λέει μια έκθεση του Μίτσιγκαν ε, του 2018. Και αυτό θα πρέπει να πούμε σε διάσημους όπως ο Λεωνάρτο Δικάπριο ή και άλλους παρόντες. Φαίνεται ότι μερικοί ε, από ε, ενδιαφέρονται περισσότερο για το κλίμα από ότι για τις πατρίδες τους. Βέβαια, σε λίγες μέρες ε, στα Ηνωμένα Έθνη θα μιλήσουμε για ένα πολιτικό θεματολόγιο που ε, αντικαθιστά την επιστήμη από ιδεολογία και μετατρέπει την προκατάληψη σε μεγάλη αλήθεια και ουσιαστικά προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του κοινού και έχουμε ταυτόχρονα πολυεθνικές που καταδικάζουν σε ανεργία εκατομμύρια Ευρωπαίους και εμποδίζουν την ανάπτυξη στην Αφρική με σύνθημα απάνθρωπο για το δικό μας τρόπο ζωής. Μιλούμε για δισεκατομμύρια ευρώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν λέμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι από τις δικές τους τσέπες θα βγουν αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαρκ Μποτεγκά. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει τώρα να ε, αποφεύγουμε την αλήθεια. Έχουμε πάρα πολλούς νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη που απαιτούν να υπάρχει μια φιλόδοξη και αποτελεσματική πολιτική του κλίματος. Όμως ε, στην ε, πραγματικότητα δεν σημειώνουμε πρόοδο, ε, δεν είμαστε ικανοποιητικά αποτελεσματικοί και γι' αυτό το λόγο εγκαταλείπουμε τους νέους στην τύχη τους. Εάν λοιπόν θέλουμε να δώσουμε μία απάντηση στην μεγαλύτερη ανισότητα και αν θέλουμε να αντιδράσουμε σε, στην έλλειψη δράσεων, θα πρέπει να πάψει να υπάρχει η πολιτική λιτότητα. Πρέπει να υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις στην υποδομή Κατά δεύτερον, πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι εκατομμυριούχοι σε ολόκληρη την Ήπειρο να καταβάλουν τους φόρους τους. Να μεριμνήσουμε γι' αυτό και αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε για τους πολίτες και για τη γη. Και τέλος, να μην υπάρχει πια αυτό το εμπόριο των ε, της ανταλλαγής εκπομπών. Οι πολυεθνικές ε, προσπορίζονται πάρα πολλά χρήματα με αυτή τη διαδικασία και μόνο έτσι θα μπορεί να σωθεί ο πλανήτης. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Κρίστιαν Σίλβιου Μπουσόη. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό ε, να επιτύχουμε τους στόχους μας για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ε, έχει σημειωθεί η πρόοδος, ε, παραδείγματος χάρη όσον αφορά το στόχο που έχει σχέση με τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Παρ' όλα αυτά υπολείπονται πάρα πολλά στο κλίμα, στην βιοπικιλότητα, στο να περιοριστεί η πείνα. Το κλίμα βεβαίως είναι το πιο σημαντικό θέμα που θα συζητηθεί και στη συνάντηση κορυφής, αλλά θέλω να επισημάνω να πιστεύω την προσοχή σα στον στόχο της χιλιτίας των υπαριθμών 10, Την μείωση των ανισοτήτων. Πολλοί τον αγνοούν το στόχο αυτό. Ε, συζητάμε για πολιτικέ υγεία, για οικονομική ανάπτυξη, για βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα δεν μπορούμε πια να συζητάμε για τι ανισότητες μόνο σε χώρες ε, ε, με χαμηλά εισοδήματα. Είναι πρόκληση και σε χώρε με μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική, αλλά το εστιάζουμε μόνο εκεί δεν θα μειώσει την ανισότητα. Πρέπει να υπάρχουν στοχευμένες πολιτικές για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο Χάβι Λόπε. ο κύριος Χάβι Λόπε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η διεθνή κοινότητα θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να μιλήσει για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα είναι μια σύνοδο κορυφή που θα πρέπει να χρησιμεύσει να αντιμετωπίσουμε μια παρούσα πρόκληση και όχι μια μελλοντική απειλή. Και θα πρέπει να περάσουμε από τη ρητορική στα έργα, από τα λόγια στα έργα. Το 2015 την υιοθετήσαμε την ρητορική, τα λόγια, στη Συμφωνία των Παρισίων για να μειώσουμε την αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια όμως ήταν τα θερμότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Επίσης έχουμε όλο και περισσότερες κλιματικές καταστροφές και θεομηνίες. Το είδαμε και στην Ισπανία με τις πλημμύρες. Επίση, δεν θα πρέπει μόνο να περάσουμε από τα λόγια στα έργα, αλλά να ζητήσουμε και να πετήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετικό ρόλο στα θέματα αυτά. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα με την οικολογική μετάβαση, με την απαλλαγή από το διοξείδιο του άνθρακα και από τη μείωση των εκπομπών. Ο στόχο ε, είναι για το 2030 40%. Θα πρέπει να έχουμε ακόμη πιο φιλόδοξου στόχου και να του υλοποιήσουμε επιπλέον. Επίση, αυτή η απαραίτητη οικολογική μετάβαση θα πρέπει να είναι και δίκαιη γιατί όπως κάθε μετασχηματισμός και στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, θα έχουμε μετασχηματισμό, ε, θα χρειαστούν επενδύσει στις υποδομές, στην κινητικότητα. Θέλουμε όμως κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλίσουμε τις ε, θέσεις απασχόλησης και να έχουμε μια διέξοδο για αυτή τη μετάβαση. Γιατί η οικολογική μετάβαση και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Έχουμε το χρόνο ακόμη, θα πρέπει όμως να ανασκοποθούμε και να περάσουμε στη δράση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μόρτεν Πέτερσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για το ακούραστο έργο του για την προώθηση της μετάβασης σε ένα πράσινο πλανήτη κατά την προηγούμενη θητεία. Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το καλοκαίρι ήταν εκλογές για το κλίμα πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξαν ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να παράγουμε έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. φτάνουμε στη Σύνοδο Κορυφής χωρίς να έχουμε φτάσει σε συμφωνία για τη φιλοδοξία που έχουμε. Το να είμαστε δηλαδή ε, κλιματικά ουδέτεροι. Αυτό πρέπει να είναι η φιλοδοξία μας και θα πρέπει να, έχουμε εμείς ηγετική θέση. Έχουμε πολλές προσδοκίες από την Επιτροπή της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Θα πρέπει να θέσουμε δεσμευτικούς στόχους για το περιβάλλον, και να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία ο Επίτροπος έχει υποστηρίξει και τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είναι από τις τελευταίες φορές που έχουμε την ευκαιρία να σας δούμε στην Ολομέλεια και συγχαρητήρια για όλα όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα και από εδώ και τώρα έχουμε επίγον έργο μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μίχαελ Μπλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στι 24 Μαΐου, λίγο πριν από τι εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκατομμύρια νέοι έκαναν απεργία για το κλίμα. Απεργούν διότι δεν λαμβάνεται μέτρα δράση. Η έκθεση για το κλίμα και οι επιστήμονε μα λένε ότι μπορούμε να μειώσουμε την αλλαγή του κλίματο σε 1,5 βαθμό. Το κύριο μήνυμα είναι ότι δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει τίποτα. Θα πάτε στη Σύνοδο κορυφή με άδεια χέρια και δεν θα γυρίσετε με νέους πλέον φιλόδοξους στόχους. Είναι αποτυχία αυτό, λυπάμαι. Και γι' αυτό την Παρασκευή αυτή εκατομμύρια και παιδιά και ενήλικοι θα απεργήσουν. Θα απεργήσουν γιατί δεν μπορέσατε να τους δώσετε αυτό που ζητούν. Ένα είναι το μήνυμά τους και θέλω να το ακούσετε. Λένε δράση για το κλίμα τώρα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ιζαμπέλα Ελένα Κλότς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, και ε, την ε, εβδομάδα αυτή τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο θα κατακλειστούν από πληροφορίε και ανταποκρίσει από τη Σύνοδο Κορυφή στη Νέα Υόρκη. Είναι προφανέ ότι η οικολογική πολιτική έχει γίνει πια κεντρικό πολιτικό κίνημα σε όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ βεβαιώνει ότι οι εκδηλώσει αυτέ και η Σύνοδο Κορυφή θα δώσουν χειρά μηνύματα και θα δημιουργήσουν έναν αγώνα δρόμου προς την κορυφή μεταξύ των χωρών ε, μελών του ΟΗΕ. Και αυτό είναι απαραίτητο για να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, των συμφωνίων των Παρισίων. Και μάλιστα ως ευρωβουλευτή από τη Σιλεσία θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά να διαλέξουμε το ρυθμό αυτής της κούρση αυτού του αγώνα δρόμου και θα πρέπει να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη που θα συμβαδίζει με την ελεγγύη προς ε, περιφερειακές και κοινωνικές ε, ομάδες που νιώθουν πολύ εντονότερα στο πετσί τους τις ε, σπευσμένες αλλαγές στις δομές. Και θα πρέπει να θυμάστε, κυρίε και κύριοι, ότι στη Νέα Υόρκη θα εκπροσωπείτε και πολίτε χωρών που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση κοινωνική και χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του. Σα παρακαλώ, μην του ξεχνάτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ντολόρης Μονσεράτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε. Το έργο που πραγματοποιείς σε ένα τόσο δύσκολο χαρτοφυλάκιο της ενέργειας και των κλιματικών αλλαγών ε, χάραξε ένα πριν και ένα μετά για όλους τους Ευρωπαίους. Εσείς ε, ήσασταν ο πρωτεργάτης κινητήριος δύναμη της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κλιματικών αλλαγών για να αφήσουμε ένα καλύτερο πλανήτη στις επερχόμενες γενιές. Η Συμφωνία των Παρισίων είχε ζωτική σημασία. Και είναι δίκαιο να πούμε ότι χωρίς τη δική σου δέσμευση και προσήλωση δεν θα την είχαμε ε, καταφέρει να ε, καταλήξουμε σε αυτή. Και σημαντικός και αξέπαινος στόχος είναι η απαλλαγή από τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα η πενταετία σου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοψίζεται σε μία και μόνο λέξη, την επιτυχία. Την επιτυχία που την υλοποιούμε μόνο χάρη σε πάθος, στον ενθουσιασμό, σε διαπραγματευτική ικανότητα και σε όραμα. Πάντα αφήνουμε το στίγμα ε, της πορείας μας και το στίγμα σου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ανεξίτηλο όπως αυτό της Λογιόλαντε Παλάσιο και ως Ισπανίδα εκ βάθους καρδίας θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Είμαστε υπερήφανοι που είχαμε ένα περίφα... έναν επίτροπο σαν και σένα και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δράσεις μας στη Σύνοδο Κορυφής της Νέας Υόρκης την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Σεπ Ντάνς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε ε, που ήμουν εγώ ε, εισηγητής για το στόχο των στόχους της χιλιετίας. Οι στόχοι αυτή τη χιλιετία είναι σημαντική για να γνωρίζουμε μέχρι το 2030 πόσο θα απέχουμε από αυτού. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν απογοητεύτηκα. Πιστεύω ότι αυτό που απογοητεύει περισσότερο είναι το σύστημα οφείλουμε να δούμε προσεκτικά το πώς ακριβώς είναι οργανωμένοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διεκδικήσουν τους στόχους της χιλιετίας. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει ευχάριστα από τα σχόλια της υποψήφιας Προέδρου ότι οι στόχοι της χιλιετίας πρέπει να διατρέξουν όλες τις γενικές διευθύνσεις. Υπάρχουν τρία σενάρια και θα είμαι απόλυτα σαφής. Μόνο το πρώτο σενάριο είναι εκείνο που θα μας οδηγεί στη θέση που πρέπει να βρισκόμαστε. Είναι το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους ε, και να έχουμε βιώσιμο μέλλον. Πρέπει, οφείλουμε να επιδείξουμε ηγετικό ρόλο. Αυτό λείπει, λείπει απεγνωσμένα στην παγκόσμια σκηνή. Να απομακρυνθούμε από την άποψη ότι οι στόχοι της χιλιετίας ε, ε, μπορούν να είναι απλώς ένα τσεκάρισμα του τι ακριβώς έχει γίνει. Κύριε Επίτροπε, είσαστε στο τέλος της θητείας σας, αλλά μην ξεχνάμε τα, τις συστημικές αποτυχίες και προσπαθήσουμε να τις διορθώσουμε κατά την επόμενη θητεία της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Βάλτερ Φλέγκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε ε, Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερος που συζητούμε σήμερα το τόσο σημαντικό και κύριε σημασία ζήτημα για το παρόν και το μέλλον μας. Όταν μιλούμε για τους στόχους μας θα πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαροι. Θα πρέπει ε, στόχος μας να είναι να γίνουμε ηγέτες παγκοσμίω ε, στον αγώνα κατά πολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Δεν θα πρέπει να αρκεστούμε σε μια δεύτερη ή τρίτη θέση. Θα πρέπει να εμεί είμαστε να γίνουμε οι πρωταθλητές παγκοσμίω. Αυτό περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από εμά και θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού ε, του 2020 ε, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη δημιουργία νέων έξυπνων αξιοπρεπών και οικολογικών θέσεων εργασίας με την τεχνολογική καινοτομία. Είμα, έχουμε ευκαιρία ε, να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Έχουμε ευκαιρία να γίνουμε πρωταθλητές παγκοσμίω στα κλιματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και θα πρέπει αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε γιατί ε, σίγουρα δεν θα πρέπει ε, να μείνουμε ουραγοί. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και γιατί η φύση μπορεί χωρίς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί χωρίς τη φύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Αλεξάνδρ Φίλιπς. Ε, κυρία, συγγνώμη, Αλεξάνδρα Φίλιπς. Ευχαριστώ. Είναι ένας αγώνας που μπορούμε να κερδίσουμε και πρέπει να κερδίσουμε, όχι για μας, αλλά για τα παιδιά μας. Εμπνεύστηκα πάρα πολύ από τους νέους, από την Κρέτα και από τους νέους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βασιζόμαστε στα παιδιά μας για να βγούμε στους δρόμους, ε, όπως τα παιδιά μας που άφησαν το σχολείο τους και ε, διέσχισαν τον Ατλαντικό για να μας κάνουν να λάβουμε μέτρα δράσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα καθήκον για το περιβάλλον και όλοι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πρέπει να μειώσουμε κατά τουλάχιστον τρει βαθμού μέχρι το τέλο του αιώνα τι εκπομπέ και θα πρέπει να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για μηδενικέ εκπομπέ μέχρι το 2030, για να έχουμε μια πραγματική πράσινη συμφωνία που θα καταπολεμήσει τι ανισότητε, τη φτώχεια θα συμμετάσχω λοιπόν στις απεργίες της Παρασκευής για να απαιτήσω για το γιο μου το ράφι και για το μέλλον όλων μας να γίνει κάτι για το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Συνάδελφος Ανιές Εφρέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού διαπιστώνουμε αβυσαλές διαφορές μεταξύ των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν και των δράσεων ε, που υλοποιήθηκαν από τις χώρες, εκ των οποίων πολλές από τις χώρες είναι και σημαντικοί ε, ε, ρηπαίνοντες. Ξεχνάει η Επιτροπή σα να αναφέρει το σημαντικό ρόλο των πόλεων για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Το ίμιση του πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο ζει σε πόλεις. Τα κτίρια είναι ενεργοβόρα. Τα συστήματα θέρμανσης παροχημένα. Κυκλοφοριακό χάο. Σε ολόκληρο τον πλανήτη οι πόλει παράγουν πάνω από 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και γι' αυτό ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών υπέδειξε το ρόλο των πόλεων ως ένα από τα σημαντικότερα πεδία δράσης. Έχω λοιπόν ένα διτό ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σκοπεύει στις 23 Σεπτεμβρίου να συμπεριλάβει και το ρόλο των πόλεων και ποιες δράσεις θα προτείνει η Επιτροπή για να δείξουμε ότι έχουμε ηγετικό ρόλο σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ δίνω το λόγο στη φίλη μας Γιούτε Γκούτελαντ, ένα μισή λεπτό. Κύριε Επίτροπε, οι εκλογές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Θα πρέπει να επιτύχουμε μια σημαντική αλλαγή. Και ο ρόλος μας είναι σημαντικός και θα πρέπει να είναι ηγετικό ρόλος για ολόκληρο τον πλανήτη. Εδώ έχουμε και ε, το ρόλο του να φέρουμε στο Κοινοβούλιο την φωνή των νέων. Η εκλεγήσα πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ότι το κλίμα θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα, όπως και η βιολογική βιοπικιλότητα θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Στη Σύνοδο κορυφή της Νέα Υόρκη θα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο για το κλίμα, και για το θεματολόγιο του 2030. Όχι με κενά λόγια, αλλά με πραγματικά έργα. Για μας, τους σοσιαλδημοκράτες, θα πρέπει να δουλέψουμε, πιστεύουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε για ένα μέλλον υπέρ του κλίματος και θα πρέπει να βάλουμε ε, τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού σαν στόχο μας. Πρέπει να δείξουμε ότι αυτές είναι οι πιο σημαντικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ε, είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη από κοινού να δείξουν στη Νέα Υόρκη ότι έχουμε την πρόθεση να υλοποιήσουμε στην πράξη αυτά τα οποία έχουμε δηλώσει. Για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά τους στόχου του Παρισιού, το θεματολόγιο του 2030 και θα παράγουμε συγκεκριμένα έργα. Στη Νέα Υόρκη μας δίνεται μια ευκαιρία δεν θα πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Πρέπει να δείξουμε ότι εμείς έχουμε τον ηγετικό ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ήπειρος και θα πρέπει να δείξουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη ότι η Ευρώπη έχει καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο σημαντικές είναι οι ευθύνες μας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γιούτα Πάολους. Έχουν περάσει περίπου τέσσερα χρόνια μετά τη Συμφωνία των Παρισίων και αποδείχθηκε ότι αυτά που αποφασίσαμε ε, το να ε, μειωθεί η θερμοκρασία κατά τουλάχιστον πέντε βαθμούς αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί εντωμεταξύ τα τέσσερα χρόνια δεν έχουν μειωθεί οι εκπομπές. Και τώρα την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη θα έχουμε τη συνάντηση κορυφής. Ζητώ συγγνώμη κύριε Κανιέτη και κύριε Ελίζα, εγώ δεν πιστεύω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει δεν πιστεύω ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Μακριά είμαστε από αυτούς. Εάν λοιπόν δούμε το τι ακριβώς έχουμε υπογράψει και γιατί έχουμε δεσμευτεί, αυτά που κάνουμε δεν φτάνουν. Η επιστήμη μας λέει και ειδικά με την, μετά την ειδική έκθεση της περασμένης χρονιάς, ε, μας λέει η επιστήμη ε, ότι μπορούμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση στην ε, εκπομπή, στην, στον περιορισμό των εκπομπών. Και αυτό περιμένω από την Επιτροπή, δηλαδή σε όλους τους τομείς να δραστηριοποιηθεί και να γνωρίζει τις επιπτώσεις στην προστασία του κλίματο στι εκπομπέ. και αυτό ε, δεν αφορά μόνο την ενεργειακή πολιτική αλλά και την πολιτική μεταφορών και την εμπορική πολιτική γιατί αυτά τα οποία πράττουμε σε μεγάλο βαθμό είναι αντιπαραγωγικά. Οδηγούν στο να αυξηθούν οι εκπομπέ και να έχουμε αποψήλωση των δασών. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση να γνωρίζουμε ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα όνειρα των νέων ανθρώπων που θα κατέβουν την Παρασκευή στου δρόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Πάουλους. Η ομιλία σας προκάλεσε ε, από τον κύριο Φούρλα μία ε, ερώτηση με τη διαδικασία της ε, μπλε κάρτας. Δηλαδή, ο συνάδελφος θα ζητήσει μία διευκρίνηση από σας με επερώτηση. Αλλά εσείς κύριε Παύλου θα πρέπει να δηλώσετε αν συμφωνείτε και δέχεστε την ερώτηση του συναδέλφου σας με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Κυρία Γιούτα Παόλους, δέχεστε την ερώτηση. One of Ένα συνάδελφό σας ζητά μια διευκρίνηση. Ερωτώ λοιπόν, θέλετε να το απαντήσετε. Ποια ήταν η ερώτηση. Η ερώτηση είναι, επαναλαμβάνει ο πρόεδρο. ένα συνάδελφό σα. ζητά με τη διαδικασία της μπλε κάρτας διευκρίνηση. Εννοείται, εννοείται, φυσικά και δέχομαι. Κύριε Φούρλα, Φούρλας, έχετε το λόγο για μισό λεπτό. Είναι στήριξη σε αυτά που λέει η συνάδελφος. Ε, ακούω πάρα πολλές φορές από όλους εδώ να λένε ότι θα πρέπει η Ευρώπη μπορούμε να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο. Δεν απλά μπορούμε, επιβάλλεται να το λάβουμε αυτό τον ε, ρόλο. Αυτή την εντολή έχουμε από του Ευρωπαίου πολίτε. Και το ερώτημα είναι πώ το αναλαμβάνουμε και πώ αναλαμβάνουμε αυτή τη ευθύνη εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ωραία να λέμε ότι πρέπει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο. Πώ μπορούμε να πιέσουμε για να αναλάβουμε αυτό τον ηγετικό ρόλο ω Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παύλος. Θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση του κύριου Φούρλα. Um, thank you very much for your... Ευχαριστώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση σας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα ε, πολύ ισχυρό ρόλο, γιατί ο δικός μας ε, ο ρόλος είναι να ε, παρακολουθούμε την Επιτροπή. Αν η Επιτροπή δεν επιδείξει αρκετή εγρήγορση, τότε θα πρέπει και εμείς να δραστηριοποιηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό είναι κάτι όπου θέλω να καλέσω όλους ε, στο Κοινοβούλιο να ασχοληθούν ε, με τα θέματα του πολιτισμού μας, να συνεργαστούμε ως ομάδες, ε, να γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, γιατί τελικά έχουμε μια κοινή υποχρέωση να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες μας. ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε την ερώτηση. Eh, Σας ευχαριστώ και η τελευταία μιλήτρια από τον κατάλογο αγορητών είναι η κυρία Εντίνα Τόθ για 1,5 λεπτό. Πρόκειται για τον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ε, πρέπει να εφαρμοστεί η Συμφωνία των Παρισίων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, γιατί οι επιπτώσεις της, ε, από την κλιματική αλλαγή δεν αφορούν μόνο την οικονομία, πρόκειται για υπαρξιακό θέμα. Και θα ήθελα να καλωσορίσω ε, την πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι ηγέτες αυτού του κόσμου. Νομίζω Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να είναι ε, υπερήφανη για τα όσα έχει επιτύχει, για την αντιμετώπιση της ε, κλιματικής αλλαγής. η ε, στόχη του 2030 είναι η πιο φιλόδοξή στόχοι. Η Ουγγαρία έχει μπορέσει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και αυτό αποδεικνύεται. Ο η αύξηση του ΑΕΠ έχει αποκοπεί από τα χρήματα για την αντιμετώπιση περιορισμού των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει μόνο κατά 2% στις εκπομπές και ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί αν όμως ε, τελικά όλες οι χώρες έχουν ε, παρεμφερείς φιλοδοξίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό χαίρομαι που ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, υπογράμμισε το ότι πρέπει να υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον του πλανήτη μας. Σας ευχαριστώ. Ε, και εδώ έχουμε μια ερώτηση με τη διαδικασία της μπλε κάρτας από τον συνάδελφο Μπενχαντίτ. Συμφωνείτε? Ο κύριος Μπενχαντίτ ζήτησε με την μπλε κάρτα δυνατότητα υποβολή ερώτηση. Το δέχεστε, κύριε Τόθ? Το δέχομαι. Ευχαριστώ. Κύριε Μπενχαντήτ, έχετε μισό λεπτό για την υποβολή τη ερώτησή σα. Ε, κοιτάξτε, η ερώτησή μου κατ' ουσίαν αφορούσε περισσότερο την κυρία Πάουλου ε, και όχι την κυρία Τόθ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση προ την κυρία Πάουλου. Ε, όχι, δυστυχώ δεν γίνεται. Πέρασε η σειρά τη. Και απάντησε σε μια ερώτηση με την μπλε κάρτα η κυρία Πάολο. Θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the τώρα. Εφτά συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους όσοι τον ζήτησαν. Αρκεί φυσικά να τηρήσετε όλοι αυστηρά και πιστά το λεπτό. Ο πρώτος συνάδελφος είναι ο κύριος Ζωάν Φεγέιρα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κλιματική δράση, όπως και στο παρελθόν οι στόχοι βιώτιμης ανάπτυξης, βρέθηκα στο επίκεντρο ε, της πολιτικής και του πολιτικού λόγου. Πέρα όμως της προπαγάνδας, πέρα της καιροσκοπίας και της ε, επιφανειακής αντιμετώπισης που πολύ συχνά γίνεται, τι μένει, δυστυχώς μένουν οι ίδιες πολιτικές, οι ίδιες πολιτικές που διακύβευσαν την βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, ειρηνική συμβίωση φύσης και ανθρώπου. Και μερικοί που κάνουν μεγαλεπίβολες υποσχέσεις που, υπο, που βάζουν την υπογραφή τους στις ε, περιβαλλοντικές συμφωνίες είναι οι ίδιοι αυτοί που οδήγησαν σε πολιτικές που κατέστρεψαν την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, που εφάρμοσαν εμπορικές και αγροτικές ε, πολιτικές που οδηγούν σε μετεγκατάσταση της παραγωγής, που πλήττουν τους πιο ασθενείς ε, συνανθρώπους μας και στερούν από πολλούς συνανθρώπους μας την ικανοποίηση ακόμη και στοιχειωδών αναγκών. Τι έγινε με τη συμφωνία, την εμπορική συμφωνία με το Μερκοσούν, εκεί λάβατε υπόψη τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τη μείωση των καυσαερίων. Γιατί ουσιαστικά προσπαθούμε να διαφυλάξουμε ένα σύστημα που δεν είναι βιώσιμο, γιατί ο καπιταλισμός μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Σπυράκη είναι η επόμενη μιλήτρια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται πράγματι της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και αυτό είναι το κεκτημένο μας, Επίτροπε Κανιέτε, στα χρόνια που ηγείστε αυτής της προσπάθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται πράγματι νομοθετικά, ηγείται και στην εφαρμογή των στόχων στα κράτη-μέλη. Αλλά προφανώς αυτό που συμβαίνει δεν αρκεί η νέα πράσινη συμφωνία που θα παρουσιάσει ο αντιπρόεδρος τίμερμανς οφείλει να λάβει υπόψη της τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ανάγκη να αλλάξει γρήγορα η προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιεί με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το νέο green deal πρέπει όμως ταυτόχρονα να στηριχθεί και σε μια νέα παγκόσμια συμμαχία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μια παγκόσμια συμμαχία προθήμων που θα περιλαμβάνει κράτη που θα περιλαμβάνει περιφέρειες και που θα έχει στόχο τη νέα βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στη χρηματοδότηση της έρευνας και τις νέες τεχνολογίες χρήματα που μπορούν να προέρθουν από το δικό μας πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από τους κρατικούς προϋπολογισμούς από τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. τα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια για όλους η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας η κυκλική δραστηριότητα στην παραγωγή και πρώτα και πάνω απ' όλα η αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου μπορούν να είναι η βάση και οι πυλώνες για τη νέα πράσινη ανάπτυξη. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μαρία Γκραπίνη έχει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Θεωρώ ότι η θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ξεκάθαρη για τα θέματα αυτά. Φυσικά θέσαμε στόχους για το 2030, για το 2050 και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναλάβει καθήκοντα εντός ολίγου θα πρέπει να υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση και να βρει τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις για να μην ε, αθετήσουμε τις υποσχέσεις μας και να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2050. Βέβαια, δεν είμαστε η περιοχή που πλέον ρηπαίνει στον πλανήτη. Υπάρχουν χώρες που ρηπαίνουν πολύ περισσότερο οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα ρηπαίνουν πολύ περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Επίση, η Σύνοδο Κορυφή θα πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσει που θα πρέπει να αναλυφθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα πρέπει να εμπλακεί πολύ περισσότερο ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στα θέματα αυτά. Και επίση ε, ελπίζουμε στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να λάβουμε υπόψη την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, ανάγκη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί χωρίς επενδύσεις, καινοτομία και έρευνα δεν θα μπορέσουμε να ελοπίσουμε τους στόχου μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Έλλη Thank Ευχαριστώ. Ε, όπως ήδη ακούσαμε την Παρασκευή, νέοι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θα βγουν στους δρόμους και θα ζητήσουν να επιταχύνουμε τα μέτρα μας κατά της κλιματικής αλλαγής. Πραγματικά μας εμπνέει ε, αυτό το οποίο κάνουν. Εμείς πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη με αυτούς που απεργούν για το κλίμα. Και πρέπει ο καθένας μας να σκεφτεί τη συμπεριφορά τη συμπεριφορά την οποία έχουμε στη ζωή μας πάνω στον πλανήτη. Και επιπλέον ως εκπρόσωποι των ψηφοφόρων μας πρέπει να ε, λάβουμε μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Το μοντέλο της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων είναι κάτι το οποίο έχουμε επεκτείνει σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουμε επιταχύνει τις ε, απαράδεκτες ανισότητες. Έχουμε την ευθύνη να δείξουμε ηγετική θέση για την ε, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να αναλάβουμε δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Η νέα πράσινη συμφωνία θα πρέπει να ερμηνευτεί στην πράξη με συγκεκριμένε πολιτικέ. Να μην γίνονται επενδύσει στα ορυκτά καύσωμα. Να μην ε, ε, ε, βοηθούμε την καταστροφή των δασών. Πρέπει τι ευθύνε μα να τι λάβουμε υπόψη και η κοινωνία και η οικονομία μα θα πρέπει να είναι αυτή την οποία πραγματικά αξίζουν τα παιδιά μα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Μίκου για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να θέτουμε στόχους και να έχουμε φιλοδοξίες δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν οι πολιτικές μας επιδεινώνουν την κατάσταση αντί να την βελτιώνουν. Το IPCC μας ζήτησε μείωση ε, κατά 50% μέχρι το 2030 και οι μειώσεις αυτές δεν είναι συμβατές με την ε, ε, επέκταση του συστήματος φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και με τις ε, εισαγωγές χιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ. Γιατί το κάνουμε, γιατί η ΣΕΛ, ένας από τους μεγαλύτερους ρηπαίνοντες στον πολίτη, έχει επιτυχές λόμπινγκ έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ιδέα ότι το φυσικό αέριο είναι πιο κατάλληλο ε, καύσιμο παρά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια έννοια που τη δημιούργησε η Shell. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε ότι οι στόχοι μας δεν πρόκειται να επιτευχθούν αν δεν αντιμετωπίσουμε τον νέο φιλελευθερισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Το λόγο έχει ο κύριος Ράνταν Κανέφ. Благодаря, господин председател. А ние всички сме... Κύριε Πρόεδρε, ανησυχούμε όλοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον τομέα του κλίματος. Ανησυχούμε για τα δάση, για τους ποταμούς, για τις θάλασσες και ανησυχούμε και βεβαίως και για, για τα τρόφιμα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώ λέμε πάρα πολλά και κάνουμε πολύ λίγα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Η δική μου η απάντηση είναι ότι καμία πολιτική δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη αν η πολιτική αυτή δεν στρέφεται προς τους ανθρώπους, αν δεν λαμβάνει υπόψη της ε, τις ανάγκες των ανθρώπων, αν δεν προστατεύει τη γεωργία και ε, εάν καταστρέφει την απασχόληση όχι μόνο στη γεωργία αλλά και στη βιομηχανία. Είναι μια πολιτική η οποία δίνει περαιτέρω κίνητρα ε, θα πρέπει να δίνει περαιτέρω κίνητρα και όχι να οδηγεί του ανθρώπου στο να εγκαταλείπουν την ύπεθρο. Χρειαζόμαστε μια πολιτική προστασία του κλίματος που θα βασίζεται στην καινοτομία και την έρευνα. Σα ευχαριστώ. Και πριν ξαναδώσω το λόγο στον Επίτροπο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του ΚΑΤΣΤΙΑΙ, το λόγο έχει ο συνάδελφος Κάρλος Σοχίνιο. Οι κλιματικές αλλαγές είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε στην ιστορία της η ανθρωπότητα. Έχουμε τεράστια πρόκληση με μετριασμού των κλιματικών αλλαγών, προσαρμογής και διαφύλαξης της βιοπικιλότητας. Αυτή η κατάσταση είναι αναφυσβήτητη, παρόλο που μερικοί την αμφισβητούν, εθελοτυφλούν μπροστά στην κατάσταση και αποσύρουν την υπογραφή τους από σημαντικέ ε, συμφωνίες για τον πλανήτη. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα τη Σύνοδο Κορυφής Νέας Υόρκης με στόχο να θαρρύνουν τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να αναβυθμίσουν τις υποσχέσεις τους για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, των αερίων του θερμοκηπίου. Ήμασταν ε, από αυτούς που έχουν πρωτοστατήσει στον αγώνα των κλιματικών αλλαγών. Και η νέα Επιτροπή έχει ενισχυμένε φιλοδοξίε. Και επίση θα έχουμε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενεργειακή Ένωση. Θέλουμε μια ισχυρή συμφωνία στον ΟΗΕ και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Η πρόκληση αυτή όμως είναι παγκόσμια. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις δράσεις μας και να συγκεκριμενοποιήσουμε το σχέδιό μας. Δεν έχουμε μόνο ένα σχέδιο κλιματικής δράσης, έχουμε 27 μεμονωμένες δράσεις, αλλά και ταυτόχρονα ένα κοινοτικό σχέδιο κλιματικής δράσης. Αυτό θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος. Ακούσατε κύριε Κανιέτε τα σχόλια των Ευρωβουλευτών. Έχετε εσείς το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή που κάναμε, που δείχνει ότι η πολιτική του κλίματο ε, ε, και ανάπτυξη βρίσκονται πραγματικά στον πυρήνα τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξεκινήσω με κάποια λόγια που είπε ο κύριο Πίτερ Λίζε. Είπε ο κύριο Πίτερ Λίζε ότι μερικέ φορέ οι Ευρωπαίοι κάνουν ε, υπερβολική αυτοκριτική. Και νομίζω ότι στην ε, Νέα Υόρκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στι προσπάθειες αυτού του Κοινοβουλίου και τη προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, έχει ένα αφήγημα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η νομοθεσία μας για την ενέργεια που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 80% περίπου ε, των ψηφισάντων, η νομοθεσία για το κλίμα ψηφίστηκε εδώ με πάνω από 78% υπερψηφισάντων. Αυτό δείχνει ευρία υποστήριξη στις προτάσεις που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Πολιτική για φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα. Ποια θα είναι τώρα λοιπόν η θέση μας στη Νέα Υόρκη. Εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε αποφασιστική συμμετοχή ε, υπέρ των στόχων που όλοι έχουν ζητήσει. Τουλάχιστον 40% ε, μείωση ε, των εκπομπών. Έχουμε τη δεσμευτική νομοθεσία που απαιτείται για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς και χάρη στη φιλοδοξία, στη φιλόδοξη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε τη δυνατότητα και να υπερβούμε τους στόχους γιατί μπορεί να φτάσουμε στο 45% της μείωσης. Έχουμε λοιπόν φιλόδοξους στόχους, δεσμευτική νομοθεσία και ισχυρή διακυβέρνηση υπό την μορφή των εθνικών σχεδίων δράσης. Κανένα άλλο φορέα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν έχει κάτι τέτοιο. Αν αλλάξει η κυβέρνηση στι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλάζει και η νομοθεσία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουν οι θητείε, αλλά η πολιτική μας παραμένει ίδια. Έχουμε λοιπόν φιλόδοξους στόχους, ισχυρή νομοθεσία και έχουμε και μια ε, προοπτική κλιματικά ουδέτερης οικονομίας μέχρι το 2050. Όταν ε, ε, λοιπόν συζητούνται αυτά τα θέματα, ε, έχω την ε, προσδοκία ότι στο Συμβούλιο Ενέργειας του Δεκεμβρίου θα περάσει αυτή η κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Και αυτή η κλιματικά ουδέτερη οικονομία είναι πολύ πιο σημαντική από τους στόχους της IPCC που ζητά κλιματική ουδετερότητα μέχρι, μετά το 2060 και πριν από το 2080. Εμείς λοιπόν θα γίνουμε η πρώτη μείζον οικονομία στον πλανήτη που θα έχουμε, μηδενικά, που θα έχουμε συγγνώμη, κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050. Και η εκλεγήσα πρόεδρος, ε, κυρία Φοντερ Λάιεν, έχει δεσμευτεί για μια πράσινη συμφωνία που θα προταθεί μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της. Και εδώ θα συμπεριλαμβάνει η νομοθεσία για το κλίμα με τους στόχους δετερότητας για το 2050. Είναι πολύ ισχυρό το αφήγημά μας και επιπλέον η εκλεγήσα πρόεδρος θέλει να μειώσει τις εκπομπές κατά 50% μέχρι το 2030 και ίσως και κατά 55%. Άρα για τη Νέα Υόρκη έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ ισχυρό και θα έχουμε και την υποστήριξη των αναπτυσσομένων χωρών. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι ότι ε, εμείς είμαστε φιλόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε φιλόδοξοι, ούτε ότι ε, θα, πραγματικά θα δώσουμε τα αναμενόμενα από εμά παραδοτέα. Θα τα παραδώσουμε όλα αυτά και σημαντικό είναι ότι θα πείσουμε και άλλους να μας οικονομήσουν. Είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητέ. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι οι δωρεέ μα προ τι αναπτυσσόμενε χώρε. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι λοιπόν για αυτά τα οποία έχουμε ήδη επιτύχει και έχουμε και μακρά πορεία μπροστά μα. Εμεί ω ηγέτε σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη τη αποτελεσματικότητα τη ενέργεια και έναντι των ορυκτών καυσίμων με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην πράσινη οικονομία. Όλα αυτά είναι θέματα στα οποία θα μα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Και έχουμε και την ευθύνη του ότι πρέπει να αναλάβουμε τον ηγετικό ρόλο, γιατί αν δεν τον αναλάβουμε εμεί, κανένα άλλο δεν θα τον αναλάβει για την κλιματική αλλαγή. Και είμαι βέβαιο ότι η νέα ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει αυτό τον ηγετικό ρόλο και είμαι βέβαιο ότι και αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσουν στην επόμενη Επιτροπή την υποστήριξη που έδωσε σε μένα. Πρέπει οι προτάσει τη Επιτροπή να βελτιώνονται από αυτό το Κοινοβούλιο και το, είμαι σίγουρο ότι το Κοινοβούλιο σα θα αυξήσει τι ε, φιλοδοξίε. Θα ήθελα τώρα να κάνω το εξή σχόλιο. Το να γίνουμε κλιματικά ουδέτερη οικονομία είναι μια οικονομική και κοινωνική επανάσταση μεγαλύτερη και από την βιομηχανική επανάσταση. Γιατί αλλάζουμε τον τρόπο παραγωγή ενέργεια, αλλάζουμε τον τρόπο θέρμανση και ψήξη, αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργία τη βιομηχανία μα. Τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία παράγει τα προϊόντα της αλλάζουμε τον τρόπο μεταφορών. Όλα αυτά αποτελούν επανάσταση. Η γεωργία θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές μεθανίου, τη χρήση λιπασμάτων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ φιλόδοξα και ο αντίκτυπος σε πολλά επίπεδα θα είναι ασύμετρος, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δίκαιη μετάβαση και γι' αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αποκτά κομβική σημασία και χαίρομαι διότι η εκλεγήσα πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις, τους τομείς και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το μεγάλο μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Συστήματος τα επόμενα χρόνια χρόνια. Φιλόδοξη στάση λοιπόν για το κλίμα και προστασία των πολιτών μας, ούτω ώστε να είναι μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. Τέλος, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μετά από το σχόλιο του κ. Φερέιρα, ο οποίος αναφέρθηκε ε, στον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών και ε, της Μερκοσούρ. Θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσει στην, πολιτική, στην εμπορική πολιτική της για να προωθεί τις δράσεις για το κλίμα στις ε, χώρες εταίρους της. Και μέχρι τώρα σε όλες τις συμφωνίες που διαπραγματευθήκαμε τα τελευταία χρόνια Τηρήσαμε αυτό το στόχο και για τον τομέα του Μερκοσούρ επίσης έχουμε βάλει περιβαλλοντικά δεσμευτικές ρήτρε και όσον αφορά τη Συμφωνία του Παρισιού περιλαμβάνεται μια ισχυρότατη δέσμευση. Κάθε συμβαλόμενο μέρος δεσμεύεται να υλοποιήσει τη Συμφωνία του Κλίματος και να τηρεί τις εθνικές ε, ε, ε, δεσμεύσεις. Όποιο λοιπόν παραβιάζει του στόχου σε σχέση με τη Συμφωνία του Παρισιού, παραβιάζει και τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Και αυτό το οποίο έχει γίνει με τη Συμφωνία του Παρισιού είναι ότι όλοι οι συμβαλόμενοι έχουν αναλάβει ισχυρέ εθνικέ συνεισφορέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ και για την ομιλία σας, αλλά και για το έργο σας και για την συνεργασία που είχατε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια της θητείας σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη Σύνοδο Κορυφής της Νέας Υόρκης της επόμενης εβδομάδας. Και μακάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατήσει την ηγετική της θέση στο παγκόσμιο πρόγραμμα εργασιών για το κλίμα. Αυτά και ολοκληρώσαμε τη σχετική συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκθεση του κυρίου Γουαλτιέρη με θέμα το διορισμό της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η υποψήφια για τη θέση αυτή είναι η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ. Και πριν κηρύξω την έναρξη της σχετικής συζήτησης, θα ήθελα να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω, για όσους το γνωρίζουν ήδη, ότι στην τρέχουσα ολομέλεια θα εφαρμόσουμε ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των ετοιμάτων για συμμετοχή στη διαδικασία Catch the και στη διαδικασία της black κάρτας. Ήδη σας ενημερώσαμε και έχετε τις οδηγίες της στέδρανά σας. Οπότε, αν θέλετε να λάβετε το λόγο είτε με την μπλε κάρτα είτε στο Catch the Eye, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κουμπί το σχετικό και να εγγραφείτε ηλεκτρονικά. Τη διαδικασίες Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ψηφοφορίας που έχετε μπροστά σας. Βέβαια, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε το έτοιμά σα με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία και την ηλεκτρονική εγγραφή. Οπότε θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την ηλεκτρονική εγγραφή ζητώντας το λόγο για το Catch ή με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Περνάμε τώρα στη δεύτερη συζήτηση της, του πρωινού. Όπως ξέρετε, η έκθεση που αποτελεί τη βάση της συζήτησή μας ήταν έκθεση που είχε αναλάβει και εκπονήσει ο πρώην συνάδελφός μας, ο κύριος Ρομπέρτο Γουαλτιέρη, που εντωμεταξύ διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας. Φυσικά το ευχόμαστε καλή τύχη και καλή επιτυχία στην άσκηση των νέων καθηκόντων του. Οπότε ο κύριος Γουαλτιέρη αντικαταστάθηκε στην εισήγηση της έκθεσης αυτής από την συνάδελφο Ιρένε Τινιάλη. Χθε, μάλιστα, η κυρία Τινιάλη ανέλαβε και την Προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, τη ΕΚΟΝ, αντικαθιστώντας και στη θέση αυτή τον συνάδελφο Ρομπέρτο Γουαλτιέρη. Τη ευχόμαστε καλή επιτυχία στην άσκηση των νέων καθηκόντων της γιατί πραγματικά η Επιτροπή ΕΚΟΝ, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είναι πάρα πολύ σημαντική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Τινιάλη, που έχει έξι λεπτά στη διάθεσή της για να μας παρουσιάσει την έκθεση του κυρίου Γαλτιέρη. Και μάλιστα μου είπε ότι θέλει να εξαντλήσει το χρόνο που έχει στην αρχική της εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με αυτή την έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζει την άποψή του ε, για τον ε, διορισμό του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ένα θεσμός ε, που έγινε πυλώνας όχι μόνο για την νομισματική πολιτική αλλά για το σύνολο της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διορισμός της Κριστίν Λαγκάρ, της πρώτης γυναίκας σε αυτό το αξίωμα, είναι από μόνο του ένα ιστορικό γεγονός ε, και συμβαίνει μόνο δύο μήνες πριν από την 20η επέτειο σε αυτήν εδώ την αίθουσα του ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα είναι πρώτα απ' όλα ένα ισχυρό οικονομικό εργαλείο. Όχι μόνο είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στην κοινή αγορά, αλλά όπως ε, πολύ συχνά επισημαίνει και ο κύριος Ντράγκη στις ε, παρεμβάσεις του, είναι η προϋπόθεση ε, για να υπάρχει ισορροπία σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο. Το ευρώ δεν είναι απλά ένα οικονομικό εργαλείο. Πάνω απ' όλα είναι ένα φιλόδοξο πολιτικό εγχείρημα. Είναι ο ακρογωνιαίος λίτος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ειρήνης, της ε, ευημερία ε, αναπόφευκτο για να στηριχθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Τα τελευταία 20 χρόνια, παρά τις ατέλειες και γενικότερα τις αδυναμίες της κοινή διακυβέρνησης, το ενιαίο νόμισμα έδειξε μία μοναδική αντοχή ακόμα και αν ε, το συγκρίνει κανείς και αν ε, το ε, εντάξει και το συγκρίνει πράγματι με παλιές ισχυρές οικονομικές κρίσεις. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Προέδρων της μέσα βεβαίως στις αρμοδιότητες τους να προστατεύσουν το ενιαίο νόμισμα με συγκεκριμένες πράξεις της νομισματικής πολιτικής αυτό συνέβαλε σημαντικά στο να προστατευτεί το ευρώ και να είναι ε, το ευρώ το νόμισμα όλων των Ευρωπαίων ε, πολιτικών. Ε, οι γραπτές απαντήσεις που έδωσε η υποψήφια όπως επίσης και η ακρόαση που έλαβε χώρα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ στις 4 Σεπτεμβρίου κατά την άποψή μου αποδεικνύουν όχι μόνο το ότι η κυρία Λαγκάρντ έχει συνειδητοποιήσει το τι την περιμένει, αλλά και το ότι είναι κατάλληλη να ε, διαδεχτεί τους ε, προκατόχους της ε, και να διαφυλάξει αυτή τη σημαντική αποστολή που της ανατίθεται. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ θεωρώ ότι τελικά θα στηρίξει την εκλογή, βέβαια, αυτό εκεί δεν τελειώνει το καθήκον μας, γιατί όπως αναφέρουν οι συνθήκες ε, και σε συμφωνία με τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις της ΕΚΤ, ε, μεταξύ άλλων, μέσα από τους νομισματικούς διαλόγους, τις αιτήσει εκθέσεις και τις γραπτές ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Και όπως πάντα θα είμαστε απαιτητικοί. Θεωρούμε ένας θεσμός ο οποίος ε, έχει ένα πολύ σημαντικό καθήκον, ο θεσμός αυτός πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Αν θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας, η σταθερότητα του ευρώ ε, δεν αρκεί από μόνη της. Πρέπει να προσθέσουμε και νέους θεσμούς, νέα εργαλεία, μια πραγματική οικονομική, ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως εξάλλου αναφέρεται και στο πρόγραμμα που παρουσίασε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Εκεί περιλαμβάνονται μέτρα για να διασφαλίζεται η πλήρη εφαρμογή του κοινωνικού κοινωνικού πυλώνα. Επίσης υπάρχουν ε, ε, αναθεωρήσεις, μέτρα αναθεώρησης για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Εμείς ε, ως συνομοθέτες είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Τινάλη. Και τώρα το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ντομπρόφσκης. Έχετε το λόγο. Mr. Chair, honorable... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Τινάλη, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Νιώθω πάντα μεγάλη τιμή κάθε φορά που συμμετέχω στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σημερινή ψηφοφορία για την υποψηφιότητα ε, Τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πολύ σημαντική, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίζει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Οι συνθήκες κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία της ΕΚΤ στην διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής. Και αυτή είναι μια αρχή που προσπίζουμε ε, ολόθερμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άλλος, ε, άλλη αποστολή της ΕΚΤ είναι η εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Η ανεξαρτησία βέβαια συμβαδίζει με τη λογοδοσία και είναι σημαντική απόδειξη των μηχανισμών της ΕΚΤ ε, που είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σημερινή συζήτηση είναι απόδειξη αυτής της διαδικασίας. Και μάλιστα είναι προφανής η επιλογή του Συμβουλίου να προτείνει την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ για τη θέση της Πρόεδρου της ΕΚΤ. Ε, συμφωνεί και η ΕΚΟΝ και το ίδιο και το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΚΤ, ότι η Χριστίνα Λαγκάρτα έχει όλα τα προσόντα και τα εφόδια για τη θέση. Και μάλιστα είναι και ένα ισχυρό μήνυμα για την ισορροπία των φίλων στην ΕΚΤ. Ε, ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο τη ΕΚΤ στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία και μάλιστα εξασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών που είναι προπόθεση για μια εύρυθμη νομισματική πολιτική. Οι δράσει τη ΕΚΤ στη διάρκεια τη οικονομική και χρηματοπιστωτικής κρίση απέτρεψαν σοβαρό αποπληθωρισμό και επέτρεψαν την ε, σταθερή οικονομική ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, έχουμε χαμηλό πληθωρισμό, κάτι που χαρακτήρισε την περίοδο μετά την κρίση και ήταν χαρακτηριστικό όλων των οικονομιών και δυστυχώ δεν άλλαξε αυτό από την ε, ΕΚΤ. Θέλουμε να και φυσικά διαρθρωτικές δαπάνες και κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική που θα συνοδεύουν τις, τα μέτρα της ΕΚΤ. Θα πρέπει έτσι να διευκολύνουμε το μετασχηματισμό που χρειάζεται για τις, οικονομικές, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους απασχολόμενους ε, στα πλαίσια της εισόδου στην ψηφιακή εποχή και απέναντι στην παγκόσμια οικονομική βεβαιότητα. Ε, και η δημοσιονομική πολιτική φυσικά θα συμβάλλει στην αύξηση ε, των επενδύσεων και στην αύξηση της ζήτησης. Όλο αυτό το τόνισε η κυρία Λαγκάρτ στην ακρόαση της ε, στην ΕΚΟΝ και συμφωνούμε απόλυτα μαζί της. Μακροπρόθεσμα ε, θα πρέπει να γίνει μια εμβάθυνση της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θέλουμε επίσης καλύτερη, καλύτερη διασύνδεση των, της Ένωσης των Κεφαλαίων Αγορών και αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ευρωζώνη. Αυτά και προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία και στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε στις ομιλίες των συναδέλφων. Η πρώτη παρέμβαση θα γίνει από τον συνάδελφο Μάρκους Φέρμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν αντικείμενο πολλών συζητήσεων τα τελευταία χρόνια ίσως δίνεται η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατευθύνει περισσότερο την πολιτική από ότι θα έπρεπε με βάση το βασικό της στόχο που είναι η σταθερότητα των τιμών. Την τελευταία εβδομάδα το πρόγραμμα αγοράς επιχειρησιακών στοιχείων ήταν άλλο ένα στοιχείο το οποίο συζητήθηκε, όπως και η μείωση των επιτοκίων και ε, Πολλοί πιστεύουν ότι ε, ξεπέρασε την εμπιστοσύνη μας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Μάριο Ντράγκη. Η Κριστίν Λαγκάρντ στην συνάντηση στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων συζήτησε όλα αυτά τα θέματα και όλοι λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία είπε για τους στόχους. Το να ανταποκριθεί στους στόχους σημαίνει ε, και ε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, θα πρέπει να σταματήσει την υπερβολικά χαλαρή νομισματική πολιτική. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ε, να διατηρήσει αυτή τη χαλαρή πολιτική. Και ε, η Κριστίν Λαγκάρντ έχει πει ότι θα είναι πολιτική τη η καλύτερη επικοινωνία για την νομισματική πολιτική. Αυτό είναι απολύτω απαραίτητο γιατί είναι υπόλογοι για τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για την καλύτερη επικοινωνία ε, η κυρία Λαγκάρτ θα πρέπει να ακούει και τις κριτικές οι οποίες γίνεται και να δρά αναλόγως. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επικεντρωθεί στο καθήκον της και οι αποφάσεις της να ανταποκρίνονται στο στόχο της. Αυτά τα έχουμε πει στην κυρία Λαγκάρτ και αυτά τις επαναλαμβάνουμε σήμερα όταν ψηφίζουμε υπέρ αυτής ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Χωνάς Φερνάντες. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Μάλιστα. Έλεγα καταρχάς ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο των Πρόψης για την παρουσία του. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ την ακρόαση με την υποψήφια Πρόεδρο της ΕΚΤ. Ήταν ικανοποιητική η παρουσία της και η ομιλία της. Η υποψήφια κυρία Λαγκάρθ Ετάχθηκε υπέρ μιας συνέχειας ε, στο έργο της ΕΚΤ και στο έργο του προκατόχου της, του κυρίου Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Ντράγκη κατάφερε να διασώσει το ευρώ σε πολύ, πολύ κρίσιμες στιγμές. Επιπλέον η υποψήφια κυρία Λαγκάρτ ε, αναθεώρησε το πλαίσιο της ε, Νομισματική πολιτική, στο πλαίσιο των συνθήκων φυσικά κύριε Φέρμπερ αλλά εντός των συνθήκων υπάρχει περιθώριο λιγμών για την αναθεώρηση ε, του τρόπου εξασφάλισης της σταθερότητα των τιμών που είναι η αποστολή μεταξύ άλλων της ΕΚΤ. Και μια και είναι και εδώ ο κύριο Τονπρόσκης θα ήθελα να τονίσω ότι χρειαζόμαστε μια δημοσιονομική πολιτική που θα συνοδεύει την νομισματική πολιτική. Αλλιώ δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το έργο μας. Σας ευχαριστώ κύριε Φερνάνδες. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Λουίς Γκαρικάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε τις ικανότητες της κυρίας Λαγκάρτ. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ την ακρόαση με την υποψήφια. Εκεί ελέγξαμε τα διαπιστευτήριά τη και πραγματικά η κυρία Λαγκάρτ πέρασε τι εξετάσει και μάλιστα με καλό βαθμό. Είμαστε εδώ και έχουμε τη σχετική συζήτηση για. όχι για να επικρίνουμε τις δράσεις της έκτα τελευταία 7 χρόνια. Το, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν το θεσμικό όργανο, το μοναδικό θεσμικό όργανο που ήταν έτοιμο να καταπολεμήσει την χρηματοπιστωτική κρίση και να δράσει για να την ανατρέψει. Μερικοί λένε ότι η ΕΚΤ ε, ε, κάνει πολλά, υπερβολικά για μερικούς. Όντως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει πολλά. Όχι γιατί το θέλει, αλλά γιατί τα κράτη-μέλη δεν ε, διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο και δεν αναλαμβάνουν τα δικά τους καθήκοντα. Όπως είπε η κυρία Λαγκάρτ στην ακρόασή της, τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Τα μισά κράτη δεν έχουν δημοσιονομικό έλλειμμα, είναι κοντά στο μηδέν, δεδομένων των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων. Έτσι τα κράτη-μέλη μπορούν να επενδύσουν στο μέλλον τους. Όχι γιατί είναι καλά ή γιατί ε, εξυπηρετούν τα άλλα κράτη, αλλά πρώτα απ' όλα εξυπηρετούν τους πολίτες τους. Ε, η πατρίδα μου η Ισπανία επίσης έχει δυνατότητα να κάνει κάτι παρά την πιο περιορισμένη οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να συνεχίσει τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στην παιδεία. Έτσι θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης μας. Και τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης μπορούν να πολλαπλασιάσουν τις ενέργειές τους. Έχουμε κολλήσει, έχουμε παραλύσει. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις συζητήσεις για, την, για το επίδομα ανεργίας, για την ασφάλεια των καταθέσεων και την εγγύηση καταθέσεων και το καθεξής. Εμείς θα υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Λαγκάρτη, πιστεύουμε ότι έχει τα εφόδια, έχει τα προσόντα, θα κάνει τη δική της αποστολή, θα την επιτελέσει στο έπακρο. Το θέμα είναι εμείς θα αναλάβουμε τα δικά μας καθήκοντα και τις δικές μας ευθύνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σβέν Κιγκόλτ. Κύριε Πρόεδρε, η όλη συζήτηση για τον διορισμό της ε, κυρίας Λαγκάρτ κατά την άποψή μου ε, είναι μια παραπλανητική συζήτηση γιατί υπάρχει σαφώς ε, ένα μήνυμα ο διορισμός της κυρίας Λαγκάρτ κατ' ουσίαν είναι η επιβεβαίωση της πολιτικής ε, του κυρίου Ντράγκη και της ε, ΕΚΤ. Η ΕΚΤ ήταν εκείνη που έσωσε το ευρώ. Χωρίς την ΕΚΤ δεν θα είχαμε πια σταθερότητα τιμών γιατί το πιο ασταθές ε, νόμισμα σημαίνει ένα νόμισμα που δεν μπορεί να προσφέρει σταθερότητα. Γι' αυτό λοιπόν οι επιθέσεις κατά της ΕΚΤ ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της, αυτές οι επιθέσεις είναι παράλογες. Ανταυτού έχουμε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάνουν σωστά τα μαθήματά τους. Και αναφέρομαι σε χώρες που έχουν να αντιμετωπίσουν ε, οικονομικά προβλήματα, χώρες οι οποίε ε, πρέπει να δώσουν όθηση στην οικονομία. Δεν τα καταφέρουν αυτά. Προβλήματα όμως έχουμε και στις χώρες με πλεονάσματα που αυτή τη στιγμή απλά αποπληρώνουν χρέη αντί να έχουν ένα περιθώριο να προωθήσουν την ανάπτυξη και μέσω των περιβαλλοντικών μέτρων. Γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ που η κυρία Λαγκάρτ είπε με απόλυτη σαφήνεια ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν μια ξεκάθαρη δημοσιονομική πολιτική. Αυτή είναι η απόλυτη προπόθεση έτσι ώστε η νομισματική πολιτική να μην αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω υπερβολική χαλαρότητα και είναι και σαφέ το μήνυμα. Πρώτη φορά ε, γυναίκα ε, πρόεδρο και πρασίνισμα τη νομισματική πολιτική. Επ' αυτόν δεσμεύτηκε η κυρία Λαγκάρτ και εμεί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Γκέρολφ Άνεμανς. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ε, πλέον τρία κόμματα τα οποία ε, είναι τα μεγαλύτερα και αποτελούν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, με τα τρίκ που κάνατε, μπορέσατε να καταφέρετε να κυριαρχήσετε στις βασικές θέσεις. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, Μακρόν, Ούρσουλα Φοντελάιν και οι Στέλε, τα πέντε αστέρια, αναγκάστηκαν να ενταχθούν ε, σε αυτή την πλειοψηφία και κάποιοι Πολωνοί από το ECR και αυτοί ψήφισαν την κυρία Φοντελάιν. ΕΚΤ, η κυρία Λαγκάρντ, ξέρουμε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει λανθασμένη πολιτική, θα εφαρμόζει την πολιτική του Ντράγκη, μεταφορά χρημάτων με ελικόπτερα, κυρίως για να μπορεί να σώσει χώρες που έχουν υπερβολικό χρέος, κρατικό χρέος. Η κυρία Λαγκάρντ, τα χειροκροτήματα για εσάς είναι όπως η ορχήστρα στον Τιτανικό. Εμείς θα καταψηφίσουμε προφανώς. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Ντέρκ Γιάνν Έπινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο πιο ισχυρός φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Βλέποντας αυτά τα οποία συμβαίνουν, βλέπουμε ότι υπάρχει διαίρεση μεταξύ των μελών, μεταξύ βορράς-νότου στην Ευρώπη, μεταξύ πολιτικών σε διάφορες χώρες, ακόμη και μεταξύ πολιτικών στην ίδια χώρα. Ο κύριος ε, Ντράγκη κρατούσε το χειρό και έλεγε ότι θα συνεχίσει να τυπώνει χρήματα, να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο χρέος δηλαδή και να έχει όσο δυνατόν χαμηλότερα επιτόκια. Κύριε Πρόεδρε, οι πρόεδροι των ε, κεντρικών τραπεζών της Ολλανδίας, της Γερμανίας και άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες ε, ξεσηκώθηκαν. 60% της ε, οικονομικής αξίας της Ευρωζώνης, της οικονομικής δηλαδή ισχύω της Ευρωζώνης, αντιτάθηκε στον κύριο Ντράγκη και παρόλα αυτά ο κύριος Ντράγκη συνέχισε την πορεία του. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη της κυρίας Λαγκάρντ, αλλά δεν είναι εδώ, είναι η πολιτική της καινής θέσης. Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα τελικά, οι καταθέτες, των οποίων η αξία των καταθέσεων μειώνεται και οι συνταξιούχοι της Ευρώπης και οι νέοι της Ευρώπης, γιατί πού πηγαίνουμε με το ευρώ. Έχουμε μια συνεχή ύφεση, οι πολίτες είναι αδύναμοι έναντι σε όλες αυτές τις δυνάμεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για δύο λεπτά κυρία Μανού Ομπρί. Αγαπητοί συνάδελφοι, τι περίεργη αίσθηση για τους νέους εκλεγέντες ευρωβουλευτές να έχουμε τη συζήτηση για τον πρόεδρο της ΕΚΤ χωρίς η μοναδική υποψήφιος η κυρία Λαγκάρτα καταδέχεται να έρθει εδώ και να μας θυμίσει με την παρουσία της. Γνωρίζουμε το ρόλο της ΕΚΤ και τους στόχους που πρέπει να επιδιώξει. Το νόμισμα έχει πολιτικό χαρακτήρα. Δεν είναι ουδέτερο ούτε για το κλίμα ούτε για τις ανισότητες. Αλλά τις ανισότητες τις γνωρίζει η κυρία Λαγκάρτ και της είχε ψωμοτήρι όταν ε, ε, διεκδικούσε την υποψηφιότητα στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, αλλά στην ε, πολιτική της τίποτα. Και όταν μιλούμε για το κλίμα και την ανισότητα, η δική της απάντηση είναι η σταθερότητα των τιμών. Πάνω από 2-3 ευρώ έχει δώσει στην αγορά η ΕΚΤ και παρόλα αυτά μόνο 10% έχει φτάσει στην πραγματική οικονομία. Το υπόλοιπο τροφοδότησε μία κερδοσκοπική υπομφόλιγα. Ακόμη και ο Μάριο Ντράγκη αναγνώρισε ότι η πολιτική του ευνόησε περισσότερο του πλουσίου. και η ελληνική τραγωδία έχει δείξει ότι η ΕΚΤ δεν ε, θέτει την πολιτική της στο συμφέρον της πλειοψηφία. Επίση, η κυρία Λαγκάρτ συμφώνησε με την κυρία Φοντελάιν για το Green Deal, για, ε, για το Οικολογικό Σύμφωνο. Θα ε, φέρουμε όμως τους ε, υπέτειους ε, ενώπιον των ευθυνών τους, τις πολυεθνικές που κυρίως ρηπαίνουν. Όχι, θα δανείσει στις χώρες για να, για να χρηματοδοτήσει την οικολογική τους μετάβαση. Όχι, θα χρηματοδοτήσει τις οικολογικές επενδύσεις. Όχι, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διαταράξουμε ή να στρεβλώσουμε την ε, πανίσχυρη αγορά, ε, την οικονομία της αγοράς. Επίσης, δεν θέλει την νομισματική ένωση να τη φέρει στην υπηρεσία της ε, οικονομικής και, νο... και κοινωνικής ισότητας. Θα πρέπει να σταματήσουμε τις ε, ρηπογόνες ενέργειες. Θα πρέπει να ε, χρηματοδοτήσουμε τις οικολογικές δράσεις και τις οικολογικές επενδύσεις. Αυτά θα θέλαμε να πούμε στην κυρία Λαγκάρτ, αν είχε καταδεχθεί να έρθει σήμερα. Και να μην συνεχίσουμε τις ενέργειες και τις συζητήσεις αυτές. Δεν έχουν νόημα έχουμε μία νομισματική πολιτική που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξυπηρετούν τον άνθρωπο και τον πλανήτη και όχι τις πολυεθνικές. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριος Νικολάου Αλαβάνος έχει το λόγο. το κεφάλαιο, η κυβερνήση κυρία Πρόεδρε, ανησυχούν για μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Προετοιμάζονται θωρακίζοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις τράπεζες, τα μεγάλα μονοπόλια που την περασμένη δεκαετία έλαβαν εκατοντάδε δισεκατομμύρια σαν ενέσει ρευστότητα χρήματα που κόβονται από τους μισθού τις συντάξει τα δικαιώματα των λαών τη Ευρώπη. η πολιτική τη τραπεζική ολοκλήρωση του δημοσιονομικού χώρου απαιτεί ξεκαθάρισμα των τραπεζών από κόκκινα δάνεια παραχωρώντα τα και σε ιδιωτικά funds εστιάζοντα του εκατοντάδε χιλιάδε μικροοφιλέτε σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση που εκβιάζονται με πληστηριασμού και κατασχέσει αντί στι τεράστιε οφειλέ των επιχειρηματιών η ανάδειξη προέδρου της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας δεν είναι ζήτημα προσώπου. η δεδομένη αντιλαϊκή αποστολή της τράπεζας της ευρωπαϊκής ένωσης δεν αλλάζει. όποιος αναλάβει θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα την ενισχυμένη υποπτία, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα ενώ τα όποια σχέδια χαλάρωση θα αφορούν και πάλι τι μεγάλε επιχειρήσει. αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα. οι λαοί τη Ευρώπη πρέπει να οργανωθούν να παλέψουν για τι σύγχρονε ανάγκε του κόντρα στο κέρδο και την εξουσία των μονοπωλίων σε κάθε χώρα. Thank ευχαριστούμε. λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην Προεδρία. Για το μεγαλύτερο μέρος ε, της ε, επαγγελματικής μου ζωής ήμουν ε, τραπεζή της Κεντρικής Τράπεζας, επομένως είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Έχουμε την τύχη να έχουμε εξαιρετικούς πρόεδρους της Κεντρικής Τράπεζας, όπως ο Jean-Claude Trichet και ο Μάριο Ντράγκη και πρέπει να κρατήσουμε τον πύχη ψηλά ελέγχθη ότι άλλαξε η Κεντρική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια. Αντί να εξετάζουμε ακαδημαϊκούς ε, ή υπεπειραμένους τραπεζίτες, αυτοί οι οποίοι ορίζονται ε, πρέπει να έχουν και ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο, αλλά να έχουν ε, και πολιτικές δεξιότητες και εμπειρία από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Από αυτή την άποψη, η Κριστίν Λαγκάρτ πιστεύω ότι είναι εξαιρετική επιλογή και θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου υποθέτω ότι υποστηρίχθηκε και στην ακρόαση στην εικόνα που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Παραμένει ένα σημαντικός κίνδυνος. Φαίνεται ότι πολλοί υπουργοί και πολιτικοί πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια μυστηριώδης μαγική πολιτική που μπορεί να υποκαταστήσει τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι η Κριστίν Λαγκάρντ είναι ενδεδειγμένη για να τονίσει τη σημασία και άλλων πολιτικών και όχι μόνο της νομισματικής πολιτικής και ελπίζω να την ακούσουν οι Υπουργοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Μαυρίδης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ. Θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα που αφορούν το μέλλον και τον δίκαιο ανταγωνισμό. Πρώτον, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων δεν οφείλεται τόσο σε τεχνικά θέματα που υπάρχουν αλλά είναι διαχειρίσιμα οφείλεται περισσότερο σε πολιτική εναντίωση από συγκεκριμένα κράτη μέλη. έχουμε δηλαδή τώρα τραπεζική ένωση χωρίς κοινή προστασία των μικροκαταθετών έχουμε κοινό σπίτι χωρίς κοινή οροφή και αυτό δεν είναι τεχνικό θέμα. τα κράτη που πλήγηκαν ιδιαίτερα από την τραπεζική κρίση αποδέχτηκαν τους δύο πρώτους πυλώνες της τραπεζικής ένωσης με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. και το δεύτερο θέμα επιπλέον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία απαιτεί την εξάλληψη των καταχρηστικών πρακτικών που δυστυχώς χρησιμοποιούνται και επιβιώνουν ιδιαίτερα λόγω της δύναμης που έχουν οι τράπεζες απέναντι στους δανειολήπτες. γι' αυτό λοιπόν αναμένουμε από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να έχει πιο ενεργητικό και δραστικό ρόλο. Thank you for one Σας ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό η κυρία Γιόν Κουρτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μας εκπλήσει το να προδικάζουμε τη μελλοντική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ θα περάσουν λίγε εβδομάδε μέχρι η νέα πρόεδρος, η κυρία Λαγκάρτ, να αναλάβει το ρόλο τη. Και γνωρίζετε ότι αν επιβεβαιωθεί σε αυτό το ρόλο τη επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να συνεργάζεται με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι 25 συνολικά, 6 μέλη του Διοικητηρίου και 19 από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Επομένως, μιλάμε για μια ε, ομαδική διακυβέρνηση η κυρία Λαγκάρτ ε, περιέγραψε το στόχο της για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει, ότι θα τηρήσει το θεσμικό πλαίσιο, ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΚΤ και θα εφαρμόσει ευελιξία και πραγματισμό για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Και από τον κύριο Φέρμπερ, από το ΕΛΚ, έγινε μια ερώτηση, ε, είπε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε περισσότερο την ε, κοινωνία των πολιτών και των νέων, να ενημερώνουμε καλύτερα την κοινή γνώμη και είπε ότι η δράση της στην ΕΚΤ θα λάβει υπόψη της και τους κινδύνους για το κλίμα, που είναι μια μακροοικονομική προτεραιότητα για την ΕΚΤ. Θα πρέπει λοιπόν ε, σιγά σιγά η ΕΚΤ να ξεφορτωθεί ε, τους ε, τίτλους εταιριών που ρηπαίνουν από το χαρτοφυλάκιό της. Υπάρχουν κάποιε βραχυπρόθεσμε προκλήσει για το ΕΚΤ. Όντω. τώρα η πολιτική επιτοκίων τη ΕΚΤ είναι πολύ χαμηλά επιτόκια και αυτό μπορεί να είναι κάπω ε, ανησυχητικό. Αλλά αυτό επιτρέπει σε πολίτε να δανείζονται καλύτερα για να αποκτήσουν ε, ένα ιδιόκτητο σπίτι, παραδείγματο χάρη. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και για του επενδυτέ που θα επενδύσουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά θα πρέπει να δείξουμε και θάρρο, γιατί για πρώτη φορά δίνουμε σε μια γυναίκα με τον πραγματισμό και την εμπειρία τη Κριστίν Λαγκάτα από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, για να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εργαστεί μαζί μα τα επόμενα χρόνια σε ένα συλλογικό πνεύμα για το όφελο των πολιτών και των επιχειρήσεών μα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Για να είμαστε δίκαιοι προς όλους, θα είμαι πιο αυστηρή τήρηση του χρόνου. Ο κύριος Φουρτασούν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη Γερμανία στο χείλο τη ύφεση, στον κίνδυνο του άτακτου Brexit, τον εμπορικό πόλεμο, να ζητούμε αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να, να αυξήσει τα επιτόκια και να μην συνεχίσει την, τις μη συμβατικέ πολιτικέ, θα ήταν πραγματική αυτοκτονία. Και επίση παραβίαση τη εντολή τη. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι πολιτικέ. Θα πρέπει να αντισταθμιστούν όμω τα αρνητικά αποτελέσματα, να μειώσουμε την ε, φούσκα των ακινήτων μακροοικονομικά μέτρα. Και επίσης να μην ε, αγοράζει ε, περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον άνθρακα. Θα πρέπει να συμβάλλει και αυτή στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αλλά όπως είπαν οι συνάδελφοι, τα μέτρα της ΕΚΤ θα πρέπει να αντισταθμιστούν με μια δημοσιονομική πολιτική. Χώρες που έχουν περιθώριο για περισσότερες δαπάνες να το κάνουν για να γιατί έχουμε και το νέο κύκλο που ξεκινά. Επίση, θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για του δημοσιονομικού κανόνε. Το ζήτησε το Ευρωπαϊκό ε, Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επίση, ε, είπαμε ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι διατάξει. Μην ε, ενδώσετε σε μια μειοψηφία κρατών μελών που αντιδρά. Θα πρέπει να υλοποιηθεί και η βούληση της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αναγκαλήθηκε. Για ένα λεπτό. Κύριος Ρενάλντο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 δεν κατόρθωσαν την ε, ρευστότητα να την μεταφέρουν στην πραγματική οικονομία. Και οι επιχειρηματίε σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν είχαν την απαραίτητη ρευστότητα. Ε, δεν, ε, ακόμα και με την εφαρμογή του, της ποσοτικής χαλάρωσης. πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι εάν οι Ευρωπαίοι έχουν άμεση πρόσβαση στις, στο η κυρία Λαγκάρντ και η Επιτροπή ΕΚΟΝ δεν μπόρεσαν να δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Ε, προφανώς ε, δεν ε, προστατεύεται το ευρώ ή κατά την άποψή μας όσον μας αφορά θα πρέπει να σας πω ότι θα καταψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you. One and a half minutes, Mr. Ευχαριστώ κύριε Βανόβερτ Φέλτ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Λαγκάρντ ε, έρχεται στην ΕΚΤ ε, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ε, την προηγούμενη Πέμπτη βιώσαμε στην ΕΚΤ ένα φοβερό θέαμα πάνω από 50% καταψήφισαν την πολιτική Ντράγκη και παρόλα αυτά και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό για την κυρία Λαγκάρτ είναι ε, το θεσμικό πλαίσιο του ευρώ. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Δεν είναι έτοιμη η Τραπεζική Ένωση, η ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, και αυτή πρέπει να προχωρήσει. Ένα τρίτο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η ΕΚΤ και η κυρία Λαγκάρτ οφείλουν να κατανοήσουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερες εξηγήσεις. Περισσότερες εξηγήσεις όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής που ακολουθείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν αυτή η πολιτική εντατικοποιήθηκε και εγώ θέλω να επισημάνω τον υψηλό κίνδυνο για τη δημοσιονομική αστάθεια. Κίνδυνος είναι ότι θα μπορούσαν να προκύψουν φούσκες. Ε, οι τράπεζες ε, έχουν δυσκολία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και με την εντατικοποίηση της πολιτικής τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. Η τρίτη παρενέργεια είναι οι επιπτώσεις ε, στους απλούς καταθέτες γιατί τελικά αυτό που στηρίζονται τι είναι, είναι εταιρείε ζόμπι όπως αποκαλούνται. Το κεφάλαιο κατανέμεται σε λανθασμένους αποδέκτες και αυτό πρέπει να Ένα λεπτό κύριο Γκουσμάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να δώσει θετική γνώμη για να αναλάβει την πιο σημαντική θέση στην οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης μη εκπρόσωπος του οικονομικού δόγματος ε, του πλήγματος και του δέους, σοκ και δέος της πολιτικής αυτής. Είδαμε τις τραγικές ε, κοινωνικές ε, συνέπειες και τις ε, αντιπαραγωγικές οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες της πολιτικής της ΕΚΤ. Και όλοι όσοι αργά ή γρήγορα κατάκριναν αυτές τις πολιτικές λιτότητες, παρόλα αυτά έκαναν θετικές δηλώσεις υπέρ της Πρόεδρου της ΕΚΤ. Βέβαια, δεν είναι ευθύνη της ε, πρόεδρου ΣΕΚΤ να απελευθερώσει τη ζώνη νερό από μια πολιτική που χρησιμοποιήσει κυρίως ε, έκτακτα μέσα οικονομικά οικονομική και νομισματική πολιτική. Σήμερα όμω έχουμε κλιματική κρίση και στο μέλλον θα έχουμε και οικονομική κρίση. Γνωρίζουμε από τη σταδιοδρομία τη ότι η Κριστίν Λαγκάρτ θα είναι μια δύναμη αντίσταση και αντίδραση στι δημοσιονομικές πολιτικές δημοσίου χαρακτήρα που θα χρειαστούμε για να δώσουμε απάντηση στην κρίση που μας περιμένει. Ευχαριστώ. Να τελειώσει η διερμηνία. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Γκιαγκιώση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ως ε, ουγγρικής καταγωγής Βέλγος οικονομολόγος ε, και όπως είπε και ένας σημαντικός οικονομολόγος, ε, ένα ενιαίο νόμισμα δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς δημοσιονομική πολιτική και χωρίς κατάλληλες πολιτικές για τους μισθούς. Όπως είπε και ο Λαφαλουσής στην έκθεσή του. Βέβαια, έχουμε τεράστιες οικονομικές ανισότητες και μαζική μετακίνηση εργατικού δυναμικού από τι χώρες περιφέρειας, χώρες του κέντρου και επίσης δημογραφική παρακμή και υψηλή ενέργεια των νέων. Αν δεν αντιμετωπίσει εκ διαρθρωτικές διαφορές, ε, δυστυχώς θα αυξηθεί το κρατικό χρέος και θα ενισχυθεί η αστάθεια του ευρώ, ενώ μια πολιτική λιτότητα θα οδηγήσει σε αντιευρωπαϊκά ε, σε αντιευρωπαϊκό αίσθημα και ευρωσκεπτικισμό. Γι' αυτό θα θέλαμε στην έκθεση προτάσεις για το πώς θα μετριάσει έκτο κίνδυνο κοινωνικής καταστροφής. Ποιες είναι οι συστάσεις πολιτικής ώστε να, να μειωθεί το μισθολογικό κενό μεταξύ παλιών και νέων χωρών μελών, μεταξύ περιφερειακών και κεντρικών χωρών μελών. Ευχαριστώ κύριο Σκάρας, για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλοί από εμά. Στι συζητήσει με την κυρία Λαγκάρτ τα τελευταία χρόνια. Είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και τώρα και στην Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων διαπιστώσαμε ότι είναι το σωστό άτομο στην κατάλληλη χρονική στιγμή, στο κατάλληλο σημείο. Χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια ανεξάρτητη νομισματική πολιτική και Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος έχει την εμπειρία, ο οποίος έχει την ηρεμία και τη συνολική ευθύνη, ο οποίος έχει την προθυμία να επικοινωνήσει, μπορεί να ε, δώσει την αιτιολόγηση των πράξεων ε, με σαφήνεια. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό ομιλητή, μια αποτελεσματική ομιλήτρια που θα διοικεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα υπερασπίζεται το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα του κόσμου, το κοινό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρώ δηλαδή. Μια επιτυχημένη νομισματική πολιτική θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και την Διαθωτική πολιτική, αλλά δεν θα την υποκαταστήσει. Τα χαμηλά επιτόκια μπορούμε να τα επικρίνουμε, αλλά δεν θα πρέπει ε, να ξεχνάμε το ρόλο μας για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται και πρέπει να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, κυρία Λαλούκ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η πρώτη μου θητεία και μου κάνει εντύπωση που δεν είναι εδώ η κυρία Λαγκάντ για να ακούσει αυτά που έχουμε να, να πούμε. Και τελικά αυτή η συζήτηση είναι διαδοχή μονολέπτων και δίλεπτων ομιλιών από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό με απογοητεύει θέλω να εκφράσω κάποιε ανησυχίε. Πρώτον, για την νομισματική πολιτική. Αν είναι απολύτω απαραίτητο να έχουμε μια γενναιόδορη νομισματική πολιτική, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι υπέρ τη κερδοσκοπίας και θα πρέπει να στραφεί προς τις πράσινες επενδύσεις για να αποφύγουμε μια νέα κρίση. Και δεν έχουμε αρκετέ εγγυησει γι' αυτό. Κάτι άλλο, η διαχείριση των κρίσεων, γιατί οκτώ χρόνια είναι μακρά χρονική περίοδος και η κυρία Λαγκάρντ δεν έλαμψε με τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Χρειαζόμαστε εγγύησεις για το πώς θα εμποδίσει μια νέα κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. One minute. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριο Σπισλάρου. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα ρουμανικά. Η υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι μόνο μια αλλαγή προσώπου. Είναι ευκαιρία να έχουμε ένα νέο πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τρία στοιχεία. Χρειαζόμαστε ένα διαφανέ τραπεζικό και νομισματικό σύστημα για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ένα σύστημα που θα δείχνει μηδενική ανοχή στην διαφθορά και θα υιοθετεί ένα νέο όραμα για τις προτεραιότητές μας, ε, την ψηφιοποίηση, τις κλιματικές αλλαγές και φυσικά την ε, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης θα πρέπει να έχουμε αυστηρές δράσεις για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένου του τρέχοντος κατακαιρματισμού. Επίσης, ε, πολλοί επιχειρηματίες έχουν αποκαρδιωθεί στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τη στήριξη των χωρών που δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωζώνης ώστε να μπορέσουν σύντομα να γίνουν μέλη σε βόμενες στα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί. Χώρες όπως η Ρουμανία θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης υποστήριξης για να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Αυτά τα σημεία θα θέλαμε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της νέας Πρόεδρου της ΕΚΤ. Ο κύριος Γιακελιούνας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Ντομπρόφσκης, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο χρωματοπιστωτικός κλάδος ε, εδώ και δεκαετίες ε, αποσταθεροποίησε την οικονομία ε, και μερικές φορές υπαγορεύει την νομισματική πολιτική. Μετά την ακρόαση και τις γραπτές απαντήσεις κυρίας Λαγκάρτ, φοβούμαι ότι δυστυχώς δεν έχει καταλάβει όλες αυτές τις επιπτώσεις η κυρία Λαγκάρτ. μαζική μόχλευση και ε, επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα, δανεισμός σε ξένα νομίσματα, στο ελβετικό φράγκο για παράδειγμα και τέτοια ενυπόθηκα δάνεια, οδήγησαν σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης ε, του καταναλωτή και στην παγκόσμια κρίση. Μερικοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε παλιότερου κινδύνου. Έχουμε και νέου κινδύνου με τι νέε χρηματοπιστωτικέ τεχνολογίε, το FinTech. Έχουμε επίση τα κρυπτονομίσματα, που δεν είναι καν νομίσματα με την παραδοσιακή έννοια. Δεν είμαι βέβαιος ότι η κυρία Λαγκάρτ αντιλαμβάνεται όλους αυτούς τους κινδύνους και όλες αυτές τις διαστάσεις. Μακάρι ε, να τα πάει καλά, μακάρι να τα πάει καλά και η ΕΚΤ, γιατί και το ΕΚΤ και οι υποπτικοί οργανισμοί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στόχο έχουν να αποτρέψουν την παγκόσμια κρίση και να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέκ για δύο λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σήμερα η Ολομέλεια θα εκλέξει την κυρία Κριστίν Λαγκάρτ ε, στη θέση της ε, Προέδρου ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πριν από δύο εβδομάδες ομολόγησε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη από το 2010 αγνόησε τους νόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κυρία Λαγκάρτ είπε μάλιστα ότι αυτό μπορεί να γίνει και στο μέλλον τέτοιου είδους ε, υπερβάσεις. Αυτό και μόνο καθιστά την κυρία Λαγκάρτ ε, την πιο ειλικρινή πολιτικό δυτικά της Πράγας. Ο προκάτοχος της κυρίας Λαγκάρτ, ο Ντραγκιαβέλη, είναι εκείνος ο οποίος ετύπωσε περισσότερο χρήμα και παραβίασε με μεγαλύτερη χαρά το δίκαιο από οποιονδήποτε άλλο και οπουδήποτε αλλού. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται λιγότερο από οποιοδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου εξαιρουμένης της Ιαπωνίας και η Ευρωζώνη ακόμα λιγότερο. Η ε, γερμανική Deutsche Bank υπολογίζει ότι η αφέμαξη των γερμανών καταθετών ανέρχεται σε 648 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί δούλεψαν σκληρά για να αποκτήσουν αυτές τις καταθέσεις και με τα χρήματα αυτά το μόνο που έγινε ήταν να πλουτίσουν περισσότερο οι μέτρη του Ντράγκη. Για το λόγο αυτό ο κύριος Ντράγκη την προηγούμενη εβδομάδα στο ετοιμοθάνατο ευρώ χορήγησε τη διπλή δόση φαρμάκου. Το ευρώ, το οποίο από το 2010 βρίσκεται στην εντατική, το γεγονός ότι το ευρώ τώρα είναι εξαρτώμενο από τη μορφήνη, αυτό δεν ενοχλεί κανένα. Γιατί ο ασθενής μέχρι να εγκαταλείψει τον κόσμο του δεν θα μπορέσει να βγει από την εντατική. Κυρία Λαγκάρτε, η ειλικρίνειά σας πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Ομολογείτε ότι παραβιάζετε τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν λειτουργείτε προς το δημόσιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κοινωνικοποιεί το κόστος ανεύθυνης κυβερνητικής πολιτικής και απληστίας του ιδιωτικού τομέα. Το ευρώ δεν είναι δημόσιο αγαθό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα υποχείριο ισχυρών οικονομικών κύκλων. Για ένα λεπτό, ο κύριος Γιουρίτσα. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. η φιλελεύθερη νομισματική πολιτική αποτρέπει τις κυβερνήσεις ε, από την εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και αν δεν έχουμε πρόσφορο οικονομικό κλίμα και αν έχουμε κανόνες ε, που δεν αποδίδουν και ο πολίτης ε, βλέπει την κατάσταση του να επιδεινώνεται, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να διορθώσουμε αυτές τις αδυναμίες. Δεν μπορούμε να επαφιόμαστε μόνο σε έναν για να κάνει το έργο σε μακροοικονομικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από την νομισματική πολιτική να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Θα πρέπει να δούμε και τι αρνητικέ επιπτώσει της νομισματικής πολιτική. Μερικέ φορέ υποσκάπτει τι οικονομίε των καταθετών. Και επίση ε, κρατάει τεχνητά στη ζωή κάποιες εταιρείες ζόμπι, ετοιμοθάνατες. Και νομίζω ότι η έκθεση ήταν πολύ καλύτερη αν ήταν πιο διαφανής και αν δημοσίευε περισσότερες πληροφορίες, ε, αμήτι τι άλλο, στο ελεκτικό συνέδριο. Θέλουμε μια μελέτη κόστος, ε, ανάλυσης κόστους ε, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόστους ωφέλους, συγγνώμη. Είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι η ηγεσία της ΕΚΤ θα τροποποιήσει την πολιτική της και θα ψηφίσω ανάλογα. Ευχαριστώ. Κύριος Πεντιτσίνη. Εμείς ε, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις ε, να έχουμε ένα λόγο για να στηρίξουμε την κυρία Λαγκάρτ. Αλλά δεν τα καταφέραμε, γιατί η κυρία Λαγκάρτ είναι συνυπεύθυνη για όλες αυτές τις πολιτικές οι οποίες οδήγησαν στην αύξηση του δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το έκανε μόνο για να σώσει τις ιδιωτικές τράπεζες, τις γερμανικές και τις γαλλικές κυρίως. Ε, αυξήθηκε λοιπόν το δημόσιο χρέος ε, και τελικά επιπλήθηκαν ε, πολιτικές λιτότητες χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές, όπως είπε ο κ. Ντομπρόφσκι. Μειώθηκαν οι, οι μισθοί, οι συντάξεις. Υπήρξε μία αναδιανομή από κάτω προς τα πάνω, οι πλούσιοι πιο πλούσιοι, οι φτωχοί πιο φτωχοί. Τώρα λοιπόν μας λένε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι κατάλαβαν οι ίδιοι ότι έκαναν λάθος, αλλά τώρα πια είναι πολύ αργά εμείς δεν θα εμπιστευτούμε την κυρία Λαγκάρτ. Πρώτα να γίνουν οι αλλαγές και μετά ενδεχομένως μπορεί και να ξανακουβεντιάσουμε. Για ένα λεπτό, κύριος Γκαρσία Μαργάγιο. Sorry, the microphone. Sorry, just one moment, your microphone. <laughs> I'm trying to, to close it. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος ότι το Συμβούλιο επέλεξε την κυρία Λαγκάρτ γιατί είναι η υποψήφια που μοιάζει περισσότερο στον Τράγκη και δεν υπήρχε άλλος καλύτερο στην αγορά. Και χαίρομαι που ε, ο κύριος Τράγκη ε, μας έσωσε γιατί δεν έχουμε μόνο επιβράδυση τη οικονομία αυτή τη στιγμή, αλλά βρισκόμαστε στο χείλο μια νέα κρίση. Και οι ε, εμπειρογνώμονε λένε δεν θα είναι κρίση ζήτηση όπω ήταν αυτή του Lehman Brothers, αλλά κρίση προσφορά λόγω γεωπολιτικών παραγόντων και αιτιών. Και εγώ θα έλεγα ABCE, Αμερική, Brexit, Κίνα και Ιράν. Αυτά είναι τα αίτια της επόμενης κρίσης. Ε, κάτι που, κάτι που μπορεί να διαταράξει τις αλυσίδες παραγωγής και να μειώσει το παγκόσμιο πλούτο. Και η απάντηση θα πρέπει να είναι με βράχη πρόθεσμα η νομισματική πολιτική που ακολούθησε ο κύριος Ντράκη και θα ακολουθήσει η κυρία Λαγκάρτ. Και χώρες όπως η Γερμανία θα πρέπει να εφαρμόσουν και αυτά ολιστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να παίξει ρόλο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριο Σούστερ για ένα λεπτό. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δέχεται όλο και μεγαλύτερη κριτική ε, αρνητικά επιτόκια και για μικρές καταθέσεις. Ε, μπορεί άραγε αυτή η χαλαρή νομισματική πολιτική να εκπληρώσει τους στόχους της ή υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Αυτά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν τους απλούς ανθρώπους. Η κυρία Λαγκάρτη είπε ότι ειπε οτι συνεχισει στην πολιτική της ΕΚΤ και εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι αυτό είναι σωστό. Αύξηση των επιτοκίων αυτή τη στιγμή έχουν ε, τα πράγματα δεν θα βοηθούσε την οικονομία, θα υπήρχε διολίστηση αναπόφευκτη σε ύφεση. Όμως και αυτό το τόνισε η κυρία Λαγκάρτ, ότι μόνη της ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να στηρίξει μακροπρόθεσμα την οικονομία και να διασφαλίσει τη σταθερότητα νομίσματος. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει επεκτατική δημοσιονομική και οικονομική πολιτική. Ε, η Γερμανία φέρει την ευθύνη. Το να υπάρχει ε, ισοσκελισμένος απόλυτα προπολογισμό, αυτό είναι λάθος. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν μια αλλαγή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος ε, Ζούμε στην Ευρωζώνη εδώ και αρκετό καιρό σε μια φάση επιτοκίων που είναι χαμηλότερα τα επιτόκια από τον πληθωρισμό. Πριν από 10 χρόνια η μείωση των επιτοκίων ε, σε περίπου 2% αυτό ήταν ενδεδειγμένο. Τώρα όμως φτάσαμε σε μια φάση αρνητικών επιτοκίων του 0,05%. Ορισμένα κράτη ε, δεν εκμεταλλεύονται όμως αυτή την ιστορική ευκαιρία. Ωραία τα λένε, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω στην ΕΚΤ του κινδύνου. Δηλαδή το ότι οι κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να ισοσκελίζουν του προπολογισμού του και οι ε, οι αποταμιευτές, οι καταθέτες ε, δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μέλλον. Υπάρχει και μία τρίτη δυνατότητα, δηλαδή να διολυστήσουμε και πάλι σε οικονομικές κρίσεις. Αυτό ισχύει παραδείγματο χάρη για τις προηγούμενες κρίσεις ε, στην Ισπανία, στην Ελλάδα. Αυτά είχαν σχέση με μία αρνητική πολιτική επιτοκίων. Γι' αυτό λοιπόν θέλω στην κυρία Λαγκάρτ να πω να έχει θάρρος, να μιλήσει με τα κράτη-μέλη και από αυτή ε, την, αυστηρή πολιτική του κυρίου Ντράγκη να ξεφύγει έστω κατά τη. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο κύριος Μπαδελά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Λαγκάρντα ανακοίνωσε ότι υπό την Προεδρία τη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι διαφανέστερη και περισσότερο προσβάσιμη στου πολίτε. Είπε ότι ο ρόλο τη ΕΚΤ είναι ε, να ασχολείται και με του πολίτε και όχι μόνο με τι αγορέ. Ωραία ομιλία για κάποιον που είναι υπέρ της, ε, του απόλυτου φιλελευθερισμού. Το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κυρία Λαγκά το αγνοεί. Αυτό είναι κακό ιονός για την έναρξη της ε, Προεδρίας της, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ήδη από την χώρα της, τη Γαλλία, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ήταν επικεφαλής ενός μεγάλου αμερικανικού δικηγορικού γραφείου. Στη συνέχεια ήταν υπεύθυνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα οι αποφάσεις λαμβάνονται κάπου αλλού μακριά από την Ευρώπη. Δεν πρόκειται για το συμφέρον του λαού, πρόκειται για το συμφέρον της παγκόσμιας ελίτ και της αγγλοσαξονικής ελίτ, την οποία υπερασπίζεται η κυρία Λαγκάρντα. Το να γίνει η κλιματική αλλαγή προτεραιότητα για την ε, ΕΚΤ ε, είναι θεμελιωδώς αντίθετο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λαός της Ευρώπης βλέπει τις επιπτώσεις, τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά στην αγοραστική του δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η μόνη κεντρική τράπεζα στον κόσμο που, μπορεί, που έχει κάνει αποκλειστική της αιμονή την καταπολέμηση ε, ε, του πληθωρισμού. Χρειάζεται ανάπτυξη των τομέων του μέλλοντος και καταπολέμηση ε, της ανεργίας. Έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα να θέσουμε στην κυρία Λαγκάτ, πολύ σημαντικά ερωτήματα και λυπούμεθα για την απουσία της. Ο κύριος Σίντσιτς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σήμερα συζητούμε εδώ για το χρηματοπιστωτικό κατεστημένο. Πριν μιλήσαμε για το πολιτικό κατεστημένο. Γιατί αποσιάζει η κυρία Λαγκάρτ. Μιλούμε για τη σημαντικότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη θέση του Διευθυντού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ελάβει τις απουσίες της. Οπότε, ε, ερωτώ το ίδιο που ρώτησε και την κυρία Φοντερ Λέιεν. Τι θα κάνει στην επόμενη οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω ότι κανένας δεν γνωρίζει την απάντηση. Είδαμε τι έκανε ως ε, επικεφαλής του Δέλτα Νιτάφ, είδαμε τι έκανε για την ε, Ελλάδα, είδαμε την πολιτική λιτότητας, είδαμε τις περικοπές της συντάξης, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει φάρμακα. Και έχουμε αυτό το φαύλο κύκλο της Ευρωζώνης που θα σκάσει όταν έρθει η επόμενη κρίση. Ε, δεν θα γίνουν όλα αυτά. Ε, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως σχετίζονται με οικονομικό σύστημα και με την ανάγκη μετάβαση σε μια οικολογική πολιτική. Αλλά θέλουμε ένα οικονομικό σύστημα για να περάσουμε στην οικολογική πολιτική. Θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε λοιπόν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιατί πριν την οικολογική μετάβαση θέλουμε μια νομισματική μετάβαση. Η Κριστίν Λαγκάρτ δεν είναι νέο άνθρωπο με νέε ιδέε. Είναι business as usual, είναι το κατεστημένο. Ε, δεν πρόκειται να υποστηρίξω κάποιον που ήταν υπέρ των μέτρων λιτότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, έχουμε χώρες ε, που ε, δεν έχουν προσχωρήσει στο Ευρώπη, στην Ουγγαρία θέλουμε να μπούμε στην Ευρωζώνη. Ε, η οικονομία μας ε, γίνεται όλο και πιο ισχυρή λόγω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 5,2%. Τέσσερις φορές παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά φτάνουν και στους ε, πολίτες, αυξάνονται οι μισθοί. Θα ήθελα να ζητήσω από τη μελλοντική πρόεδρο της ΕΚΤ να εφαρμόζει νομισματικές πολιτικές που θα λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα και των χωρών της Ευρωζώνης και αυτών εκτός Ευρωζώνης. Ε, ε, όταν γίνεται κάτι στην Ευρωζώνη επηρεάζει και αυτές που είναι εκτός Ευρωζώνης. Ε, ε, αυτό ισχύει παραδείγματο χάρη για του προπολογισμού. Η νέα πρόεδρος ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη ότι ο προπολογισμό δεν θα πρέπει να βασίζεται σε πόρους από χώρε εκτός Ευρωζώνη. Τέλο, εμεί ε, θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να αλλάζουν συνεχώ οι προποθέσει για να μπορεί κανεί να προσχωρήσει στην Ευρωζώνη. Ο κύριο Μπέλκα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ ε, φροντίζει για την Ευρώπη. Ο κύριος Ντράγκη το διευκρίνησε αυτό το 2012. Το ευρώ μαζί με, το, την, ε, με την κοινή αγορά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, το πιο ε, μεγάλο ατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρώ δεν είναι μόνο υποχρέωση και ένας περιορισμός της εθνικής πολιτικής, αλλά και είναι τεράστιο ατού, ένα τεράστιο πλεονέκτημα για να παραφράσουμε ένα, μια αντίστοιχη φράση για το, ευρωπαϊκό, για το αμερικανικό δολάριο. Είναι ένα παγκόσμιο νόμισμα πια και ε, δεν θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να ανησυχούν για κρίση ρευστότητα σε, περίπτωση κρίσης. Ε, δεν χρειάζονται εθνικούς πόρους ε, και να συγκεντρώνουν από θέματα σε συνάλλαγμα. Αυτά είναι δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Αυτό θα πρέπει να το επιθυμίσουμε και στους ηθήνοντε πολιτική και στο κοινό. Και σίγουρα οι επικοινωνιακέ ικανότητε της κυρίας Λαγκάρτ θα χρησιμοποιηθούν και απέναντι στις χώρες εκτός τη Ευρωζώνης, όπως η Πολωνία. Θα ήθελα να της ευχηθώ καλή τύχη στη, στα νέα της καθήκοντα και να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξή μου προ το πρόσωπο τη κυρία Λαγκάρτ. Κύριε Πρόεδρε, ε, η πολιτική του κύριου Ντράγκη είναι τραγική. Έχουμε κυβερνήσει που πήραν φτηνό χρήμα και αυξήθηκαν κατά πολύ τιμέ των ακινήτων. Ποιο τα πλήρωσε, ο μικρό καταθέτης, τα χρήματά του δεν αξίζουν πια τίποτα. Δεν παίρνει πια επιτόκου. και μόνο αυτό φοβάται ότι έχει να αντιμετωπίσει ε, και αρνητικά επιτόκια για να τιμωρηθεί για το ότι δεν θέλει να καταναλώσει. Και τι προκύπτει τώρα, έχουμε την lame duck, την κυρία Μέρκελ, τον ε, κύριο Μακρόν που αυξάνει το δημόσιο χρέο ε, και ενδιάμεσα την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αρχίζει και διερωτάται ποιος θα πάρει την, την ΕΚΤ. Αυτή λοιπόν είναι μια βρώμικη διαπραγμάτευση. Ε, όποιος ε, αποταμιεύει χάνει, όποιο κάνει σωστού προπολογισμού είναι βλάκας. Η κυρία Λαγκάρτ είπε στην Επιτροπή ότι ε, δεν αποκλείεται να καταργηθεί το ρευστό και να υπάρχουν αρνητικά επιτρόκια. Εγώ αυτό το βρίσκω πολύ επικίνδυνο. Και αν δεν υπάρχουν ε, χρήματα που να μπορεί κανεί να κρύψει, ξέρετε τι θα κάνει τότε. Θα προβεί σε απαλωτριώσει σε κάτι που η κυρία Λαγκάρτ το είχε ζητήσει και παλαιότερα. Εγώ τρέμω, φοβάμαι με όλα αυτά που ακούω. Ένα λεπτό, Κύριο Κίρτσο, παρακαλώ. Στηρίζουμε την κυρία Λαγκάρντ και περιμένουμε να μα στηρίξει και αυτή, την ελληνική οικονομία δηλαδή. Θεωρούμε θετική την δήλωση που έκανε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για μελλοντική μείωση των ελληνικών πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό θα βοηθήσει την οικονομία μας να λειτουργήσει καλύτερα. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μας βοηθήσει στην πιο γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων, των non-performing loans. Ε, νομίζω και ο κύριος Ενρία του SSM πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση και στηριζόμαστε σε αυτούς για να βοηθηθούν οι τράπεζες οι ελληνικές που έχουν πρόβλημα και η πραγματική οικονομία. Επομένως, η κυρία Λαγκάρτ μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κάνει πολλά για την ελληνική οικονομία και το τρίτο που περιμένουμε είναι να μας βάλει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που δυστυχώς χάσαμε με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης την περίοδο Ντράγκη αλλά βέβαια για να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που συνεχίζεται θα πρέπει τα ελληνικά ομόλογα να πάρουν επενδυτική βαθμίδα. Αυτό ακριβώς θα επιδιώξουμε. Όσο καλύτερα πάει η ελληνική οικονομία, τόσο το καλύτερο για την Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα για ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Obrigado. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ προφανώς έχει τα προσόντα και την προσωπική και πολιτική εμπειρία για να γίνει πρόεδρος της ΕΚΤ. Και για τρεις λόγους κυρίως θα την υπερψηφίσουμε οι σοσιαλιστές. Καταρχήν, γιατί είναι υπέρ της συνέχιση της νομισματικής πολιτικής του Μάριο Ντράγκη και εμείς χρειαζόμαστε ως επικεφαλής του ΕΚΤ κάποιον που θα είναι ε, έτοιμος να κατανικήσει τις αντιστάσεις και να κάνει ό,τι χρειάζεται για να, να διασώσει το ευρώ ακόμη και μια μη συμβατική νομισματική πολιτική. Δεύτερον, θα την υπερψηφίσουμε γιατί είναι υπέρ μια δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, πιο φιλική προ ε, την ανάπτυξη. Και επίση είναι υπέρ τη μεταρρύθμιση τη ΩΝΕ, υπέρ τη δημιουργία τη Τραπεζική Ένωση και τη ενίσχυση τη δημοκρατική νομοποίηση τη οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μας υποσχέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Λαγκάρτ και αυτά θα απαιτήσουμε να τηρήσει στη θητεία της. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο Σάντ. Προσθέτω και εγώ τη φωνή μου σε αυτούς που υποστηρίζουν ε, την κυρία Λαγκάρτ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρότι δεν συμφωνώ με όλα τα στοιχεία από το ε, πολιτικό της ε, παρελθόν. Η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Παρ' όλα αυτά θέλω να υποστηρίξω κάτι το οποίο το ξεχνάμε συνήθως Μιλάμε για τις μικρές ε, ε, τράπεζες της ε, Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης και τις Ευρωπαϊκές και τις Κεντρικές Τράπεζες των Ευρωπαϊκών χωρών. Ξεχνάμε το ότι χρειάζονται υποστήριξη μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη που προσπαθούν να βρουν κεφάλαιο. Αυτές οι τράπεζες έχουν παραβλεφθεί γιατί δεν έχει ε, ακολουθηθεί διαφορετική στάση για αυτές συγκεκριμένα και αυτό είναι ένα πρόβλημα, Θα θεωρήσουμε ίσονο σημασία. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από τον επόμενο μιλητή. Ξέχασα την κυρία Φιτζέραλντ που ήταν στον κατάλογο των ομιλητών. Σας δίνω το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν χαιρετίζω την, τον, τον διορισμό της κυρίας Λαγκάρτ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα έχουμε τώρα μια ε, γυναίκα και, στο Ευρωπαϊκό, και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γυναίκες σε δύο σημαντικούς φορείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί πρόοδο για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο πολύ συγκεκριμένου ε, και σημαντικού τομεί. Η κυρία Λαγκάτ στην Επιτροπή Οίκων ε, τόνισε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να καταλάβει το ρόλο τη και να τον εξηγήσει όχι μόνο στι αγορέ αλλά και στου πολίτε. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια κατευθυντήρια γραμμή για την ΕΚΤ. Θα πρέπει δηλαδή να ακούει τη φωνή των πολιτών. Η εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα είναι κάτω από το 50% από το 2008 και μετά και αυτό είναι δείγμα του ότι μετά την οικονομική κρίση πλήττεται η δημοσιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ιρλανδία είχαμε σαφώς αυτό το φαινόμενο και παραμένει μέχρι τώρα. Ε, το τραπεζικό μα σύστημα είναι πολύ συγκεντρωτικό με μικρό εξωτερικό ανταγωνισμό και αντιμετωπίζουμε και τι προκλήσει του Brexit. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εκφράζω την εκτίμησή μου για την κυρία Λαγκάρτ ε, για την βοήθεια που έδωσε στην Ιρλανδία τα δύσκολα χρόνια τη οικονομική κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. 1,5 λεπτό, κυρία Ντελάνγκε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι διάφορες απόψεις που ακούγονται δείχνουν καταρχήν τις τεράστιες προκλήσεις που περιμένουν την Χριστίν Λαγκάρντ. 19 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και 27-28 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με οικονομίες οι οποίες αποκλίνουν και η κυρία Λαγκάρντ θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει ευρωπαϊκές λύσεις για όλους. Ε, δεύτερον, πολύ σωστά έχουμε επιλέξει μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που να μην διοικείται από πολιτικούς. Βέβαια, οι δευτερεύουσες συνέπειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, σαφώς έχουν επιπτώσεις σε αυτούς οι οποίοι έχουν ε, κάποιες οικονομίες τις οποίες έχουν καταθέσει για τα γυρατιά τους ή για τα παιδιά τους. Αυτά λοιπόν, ε, τα, αυτές τις δευτερογενείς επιπτώσεις πρέπει να τις λάβει ε, υπόψη η κυρία Λαγκάρντα. Κάνω λοιπόν μια έκκληση στη σημερινή συζήτηση να λάβουμε υπόψη και τις δευτερογενείς επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά ταμεία. Μιλάμε για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ποιος είναι αυτός ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής? Ε, είναι το να έχουμε χρέη και τα χρέη μας να τα μεταφέρουμε στις νέες γενιές ή είναι να σεβόμαστε και τις μεσαίες τάξεις που προσπαθούν να εξοικονομήσουν και να αποταμιεύσουν χρήματα για τα γυρατιά τους. Πιστεύω το δεύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye και σας ευχαριστώ που λάβατε μέρος ε, στην ηλεκτρονική δοκιμή που κάναμε. Εφτά δήλωσαν ε, ενδιαφέρον να μιλήσουν. Θα τους ε, δώσω το λόγο σε όλους. Ο κύριος Βαντάλεν πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το βασικό για τον Πρόεδρο της ΕΚΤ είναι τι πολιτική θα ασκήσει. Πριν από 7 χρόνια η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνέβαλε στην αντιμετώπιση ή μάλλον συνέβαλε στην κρίση τη χρηματοπιστωτική και συνέχισε την πολιτική της παρά την έλευση της χρηματοπιστωτικής κρίσης δισεκατομμύρια ευρώ δώστηκα, δόθηκαν για να σωθούν χώρες και δυστυχώς ο, ε, ο κύριος Ντράγκη ενίσχυσε αυτή την πολιτική. Ευτυχώς φεύγει τώρα. Φθήν το χρήμα με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια και οι συνταξιούχοι δεινοπαθούν. Οι καταθέτες έχασαν τις οικονομίες τους και σε πολλές χώρες Ευρωζώνης ε, δεν έγιναν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ο πρόεδρος της ε, Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας αντέδρασαν. Αντέδρασε μαζί με άλλου συναδέλφου του. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική και ελπίζω να ανατρέψει την τάση η κυρία Λαγκάρτ. Κλείσαμε το κατάλογο με το Catch the Eye. Δύο ακόμη προσθέθηκα στο, στο κατάλογο και τελειώνουμε. Ο κύριος Μάρκες. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αντίθετα από την θέση ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η κυρία Λαγκάρτ υποσχέθηκε ότι θα διατηρήσει την τρέχουσα νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, κυρίως τα μη παραδοσιακά εργαλεία, τα οποία υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια και μάλιστα και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή η πολιτική έσωσε το ευρώ και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να πάμε πίσω. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε το διορισμό της ε, κυρίας ε, Λαγκάρκ, αλλά σας προειδοποιώ, εάν τα γεράκια του μονεταρισμού αρχίσουν να δαγκώνουν, τότε ε, πρέπει να ξέρετε την πρώτη που θα δαγκώσουν θα είναι την ΕΚΤ. Εμείς χρειαζόμαστε μια νομισματική πολιτική σαν αυτή που είχαμε από το 2014. Βέβαια, όπως ανέφερε και η υποψήφια, έχει φτάσει πλέον η στιγμή και η δημοσιονομική πολιτική να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Χώρε με μακροοικονομικά ε, πλεονάσματα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να έχουμε σταθερή οικονομία. Μακροπρόθεσμα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση. Διακόπτει η πρόεδρος ε, το ομιλητή και λέει στον ομιλητή ένα λεπτό είχατε. Επόμενο ερωτών, παρεμβαίνων. Κύριος Γιούρκη.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 ε, θέλω να πω το εξή. Ε, οι υπεύθυνοι πολιτικοί ε, πρέπει να σταματήσουν να βρίζουν το ευρώ. Ε, το ευρώ είναι πολύ καλύτερο από ό,τι πιστεύουν πολλοί. στο σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο ευρώ. Η κυρία Λαγκάρντ, εγώ σας λέω, ε, και σας καλώ να μην ε, συνεχίσετε την πολιτική του κυρίου Ντράγκη. Αυτό πρέπει ε, να το κατανοούν όλοι γιατί θα δημιουργηθούν νέες φούσκες καταναλωτικές που θα τις φορτώσουμε στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό λοιπόν η κυρία Λαγκάρτ λέει ότι αυτή θα συνεχίσει αυτή την πολιτική. Εμείς όμως πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται έτσι ώστε να πετύχουμε την απομάκρυνση από την τρέχουσα νομισματική πολιτική. Να στηρίξουμε τους καταθέτες, όχι τους οφειλέτες. Να βρούμε μία ισορροπία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, κύριος Φερέιρα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ΕΚΤ το ΔΝΤ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκαναν μια τρόικα που επενέβη στην Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Η κυρία Λαγκάρτ, ε, η υποψήφια για τη θέση της Προεδρίας της ΕΚΤ, ήταν υπέρ της ε, ε επεκτατικής λιτότητας που ενέπρευσε το πρόγραμμα της Τρόικα. Ήταν ε, τραγικά από οικονομική και κοινωνική άποψη τα αποτελέσματα της επέμβασης Τρόικα. Και τώρα... συνέβαλε στην πολιτική αυτή ε, αναγνώρισε κάποια λάθη βέβαια η κυρία Λαγκάρτα, αλλά δεν άλλαξε τις πεπιθήσεις της. Ε, και μάλιστα πρόσφατα συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απείλησε την Πορτογαλία να μην χαλαρώσει τη δημοσιονομική της πολιτική, ε, στηρίζοντας τις δημοσιονομικές και δημοσιονομικούς περιορισμούς. Και τώρα αυτή η υποψήφια έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δεξιά, οι σοσιαλιστές, ακόμη και οι πράσινοι τη στηρίζουν. Είμαστε βέβαια στην επόμενη κρίση της Ευρωζώνης ε, θα δουν οι υποστηρικτές της Λαγκάρτη θα γίνει. Νομίζω ότι η μισθή και η απασχόληση θα είναι οι σταθεροποιητικοί παράγοντες. Ο πρόεδρος διακόπτη, περάσατε το λεπτό σας ε, κύριε Φεραίρα. Λυπούμε πολύ, αλλά δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Προσπαθώ να είμαι δίκαιη απέναντι στους συναδέλφους κύριε Πρόεδρε, οπότε ένα λεπτό προβλέπετε για το Κατσδιά. Κύριε Μπόκοβιτς, είμαι σίγουρη ότι δεν θα με απογοητεύσετε. Σας ευχαριστώ. Το ευρώ είναι το ισχυρό οικονομικό νόμισμα που χρησιμοποιούν 330 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σε 19 χώρες. Είναι ένα νόμισμα που καλύπτει το 16,9% του παγκόσμιου ΑΕΠ και 30% του παγκόσμιου εμπορίου. Ε, Πέραν από ένα ισχυρό ευρώ όμω, χρειαζόμαστε και κάποιε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει στι διάφορε χώρε, ώστε να εξασφαλίσουμε σταθερέ οικονομικά και κοινωνικά πολιτικέ, για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ευστάθεια στου πολίτε. Θέλουμε και στιβαρά και στεναρά τραπεζικά συστήματα, ανθεκτικά και να μην είναι έρμεα των κόκκινων δανείων που επεκτάθηκαν στη διάρκεια της κρίσης. Η ΕΚΤ συνέβαλε στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία να ξεπεράσουν οι χώρες αυτές την τραπεζική κρίση και ακόμη και σε περίπτωση κρίσης η ΕΚΤ βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι πολύ πεπειραμένη επαγγελματία η κυρία Λαγκάρτ και θα την υπερψηφίσω και εγώ σήμερα. Κύριος Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές οικονομικές προκλήσεις και παράλληλα βλέπουμε ότι η νομισματική πολιτική έχει όρια. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε κατά νου, δεν πρέπει να είμαστε σαν τον Τραμπ, που λέει ότι αν η Federal Reserve κάνει λάθος, τότε αυτό σημαίνει ότι λάθος κάνει όλη η χώρα. Μέχρι τώρα βέβαια το πρόγραμμα της ΕΚΤ ίσως ε, να μην ήταν τόσο καλό όσο το θέλαμε. Είδαμε ότι υπάρχουν άλλα συστήματα τα οποία έχουν λιγότερες επιπτώσεις. Αυτό το διαπίστωσε ήδη ο Κέινς. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το πώς μπορούμε να συντονίζουμε σωστά τη νομισματική πολιτική. Βεβαίως και δεν πρέπει να είμαστε αντιπαραγωγικοί με την νομισματική πολιτική. Οφείλουμε σε μία φάση ύφεση ε, να αναζητούμε μία νομισματική πολιτική που να συμβαδίζει με την πολιτική του χρήματο και να είναι καλή για το σύνολο τη Ευρώπη. Τα θέματα του κλίματο, τα οικονομικά, τα προβλήματα τη μετανάστευση, όλα αυτά απαιτούν ε, περισσότερη και όχι λιγότερη συνεργασία. Ο κ. Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να εκφράσω την ε, λύπη της ευρωομάδας της αριστεράς γιατί η κυρία λαγκάρντ σήμερα αποφάσισε να απουσιάσει να σνομπάρει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. ίσως είναι συνηθισμένη από τον τρόπο που λειτουργούσε ως επικεφαλής του διεθνούς νομισματικού ταμείου αλλά εδώ η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα οφείλει να ενισχύσει τη δημοκρατική λογοδοσία δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την κυρία Λαγκάρτ, ως ευρωομάδα της Αριστεράς δεν θα την ψηφίσουμε, γιατί είμαστε αντίθετοι με τις συνταγές που εφάρμοσε ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε χώρες όπως η Ελλάδα, που προκάλεσαν απίστευτη ύφεση, τριπλάσια ενεργεία, τεράστιο κοινωνικό πόνο. Και δεν έχουμε πιστεί ότι θα εφαρμόσει θετικές πολιτικές. Είναι όμως αλήθεια ότι εκτός από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η ώρα και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική υπέρ της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Mr. Polchak, minute. Ο ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω το διορισμό της κυρίας Λαγκάντο σε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι είναι μια πεπειραμένη πολιτικός. Και για μένα κέρια σημασία έχει το ότι υποστηρίζει την ολοκλήρωση της Νομισματικής Ένωσης και επίσης το ότι θέλει να εξηγήσει τη νομισματική πολιτική στους πολίτες. Πιστεύω ότι πρέπει οι πολίτες της Ευρώπης να γνωρίζουν τις πολιτικές μας. Μπορεί να μην έχει η Τσεχία το ευρώ, αλλά πιστεύω ότι το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα. Και η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να υποστηρίξει την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα χρειαζόμαστε σταθερότητα στο σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποίησε αντισυμβατικά μέτρα στο παρελθόν για να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική και υπό την Κριστίν Λαγκάρντ. Υποστηρίζω λοιπόν το διορισμό τη και από τη συζήτηση νομίζω φαίνεται ότι οι περισσότεροι την υποστηρίζουν. Ευχαριστώ. Γκραπίνη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ΕΚΤ βεβαίως είναι σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη και για την σταθερότητα του νομίσματος. Η κυρία Λαγκάρντ έχει την απαραίτητη κατάρτιση και έχει δείξει ότι έχει τις ικανότητες για τη θέση. Και εγώ και ορισμένοι συνάδελφοι έχουν επικρίνει την ΕΚΤ για τις πολιτικές που ακολούθησε κάποια στιγμή. Συμφωνώ ότι η κυρία Λαγκάρντ τώρα αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Η χώρα μου δεν είναι μέρος της Ευρωζώνης καταλαβαίνω ότι ενδέχεται να υπάρχουν νέε οικονομικέ κρίσει στο μέλλον και δεν πρέπει να χωρίζουμε την Ευρώπη σε ευρωζώνη και χώρε εκτό Ευρωζώνη. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλου του πολίτε και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και να είμαστε υπέρ μια πολιτικής που δεν θα οδηγεί σε αρνητικά επιτόκια. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος. Ε, κύριε Επίτροπε, βλέπετε ότι έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν οι συνάδελφοι για να ψηφίσουν. Σα δίνω το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή δεν συμμετέχει στη διαδικασία διορισμού του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρ' όλα αυτά, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διαδικασία αυτή και γι' αυτό άκουσα πολύ προσεκτικά τις απόψεις σας για την μακροοικονομική πολιτική στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε διότι το Συμβούλιο, θα θέλουμε το Συμβούλιο ε, να ορίσει ένα άτομο που θα είναι το κατάλληλο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χαιρόμαστε γιατί για πρώτη φορά πρόκειται για μια γυναίκα. Ε, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Επίτροπε, αλλά για τους συναδέλφους που μόλις μπήκαν στην Ολομέλεια, παρακαλώ να φτάσετε στις θέσεις σας ε, με ησυχία για να αφήσουμε τον Επίτροπο να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. νέο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει δύσκολο έργο και τώρα σύντομα και στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Στο άμεσο μέλλον, σε περίπτωση παρέμβαση τη ΕΚΤ απαιτείται για να απευθυνθεί μια ύφεση στι οικονομικέ δραστηριότητε. Συμμεριζόμαστε αυτό που είπε και στην Λαγκάρτ κατά την ακροασή τη. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχει ε, μπορούμε να βελτιώσουμε την όλη προσέγγιση, να υπάρξει καλύτερη υποστήριξη διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και των διαφόρων δημοσιονομικών πολιτικών. Επίση, πιστεύουμε κι εμεί. Λυπάμαι, κύριε Επίτροπε, λέει η πρόεδρο. Λυπάμαι, κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι, δεν θέλω να κατονομάσω κανέναν. Δεν σας ξέρω κι όλους με το όνομά σα. Παρακαλώ, συνάδελφοι στα δεξιά μου. Εκεί δεξιά. Λυπάμαι, λυπάμαι. Δεν θα λέω ησυχία, ησυχία, διότι δεν είμαι στη Βουλή των Κοινοτήτων να λέω order, order. Θα μου άρεσε να έχω την ίδια φωνή και επιρροή με τον πρόεδρο τη Επιτροπή των Κοινοτήτων. Ησυχία, παρακαλώ. Ο Επίτροπο Ντομπρόφσκη απαντά σε αυτά που συζητήσαμε. Δεν θα ξαναρχίσει η συζήτηση εκτό αν επικρατήσει ησυχία. Παρακαλώ, εστέ ήσυχοι, συνάδελφοι. να περιμένουμε. Δεν αρκεί η ησυχία που έχουμε τώρα. Πιστεύουμε και εμεί λέει ο επίτροπο ότι η εμβάθυνση οικονομικής νομισματικής ένωσης θα είναι υποφελή για τη λειτουργία τη Ευρωζώνης, θα είναι πιο ανθεκτική και θα προωθηθεί και η θέση του ευρώ στην παγκόσμια κλίμακα. Στην Επιτροπή για τα Οικονομικά νομισματικά Θέματα, όταν έγινε ακρόση για την Κριστίν Λαγκάρντ, είδαμε εκεί ότι το Κοινοβούλιο έχει την ίδια προσέγγιση. Ελπίζω ότι αυτή η ευθυγράμμιση απόψεων θα ανοίξει το δρόμο για να συνεχιστεί η έξοχη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, σεβόμενοι πλήρως τους αντίστοιχους ρόλους υπό την Προεδρία της ΕΚΤ από την Κριστίν Λαγκάρντ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την αντοχή σας. Πέρα στις συζητήσεις προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, έχω να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, σύμφωνα με τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη που εγκρίθηκε χτες, ο πρόεδρος προτείνει την Τετάρτη το απόγευμα η συνεδρίαση να παραταθεί μέχρι την Ενάτη βραδινή για να μπορέσουμε να μοιράσουμε σωστά τα θέματα. Ε, διαφωνείτε? Αν όχι, εγκρίνεται λοιπόν αυτή η τροποποίηση της ημέρης της διάταξης. Δεύτερη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες Ιταλικές αρχές ενημέρωσαν τον Πρόεδρο για την εκλογή του κυρίου Νικολά Ντάντι, παλιό μέλος, γνωστό συνάδελφος. Ε, εκλέγεται Ευρωβουλευτής από η Ενάτου 2019. Ο κύριος Ντάντι αντικαθιστά τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, ο οποίος όπως γνωρίζουμε ανέλαβε υπουργός στην Ιταλική κυβέρνηση. Καλωσορίζω τον νέο συνάδελφο και καλό φίλο μπορώ να πω, Ντάντι. Και θυμίζω, ο κύριος Ντάντι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός, συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των οργάνων του Κοινοβουλίου. Καλωσορίσατε θερμά κύριε Ντάντι και ε, ό,τι καλύτερο και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Er Μπορείτε να σηκωθείτε κιόλα, κύριε Ντάντι. Γεια σα. καλώς ορίσατε θερμά και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, καλή τύχη. Περνάμε λοιπόν στι ψηφοφορίε που σήμερα είναι πολύ σύντομέ χωρίς αυτό σημαίνει ότι είναι και λιγότερο σημαντικέ. Η πρώτη ψηφοφορία είναι ο διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα, τη Προέδρου, εν προκειμένου, της κυρίας Κριστίν ε, Λαγκάρτ.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 Die Abstimmung ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 394 ψήφοι υπέρ, 206 ψήφοι κατά, 49 αποχές. Συγχαρητήρια. Κυρία Λαγκάρτ. Δεύτερη ψηφοφορία διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου ε, της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται για τον Ιβ Μέρς. Επίσης μυστική ψηφοφορία άρχεται τώρα. Die Πέρας. 379 υπέρ, 230 κατά, 69 αποχές. Συγκέντρωσε λοιπόν την απαραίτητη πλειοψηφία ο κύριος Μέρους και εκλέγεται. Συγχαρητήρια. Και ε, περνούμε στην τρίτη ε, ψηφοφορία. Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία είναι η έκθεση Λόπες Αγγιλάρ. Μυστική, όχι, όχι, δεν είναι μυστική ψηφοφορία, διορθώνει ο πρόεδρος, είναι ονομαστική όμως. Αρχίζει τώρα. Πέρας. ...588 υπέρ, 59 κατά, 29 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Κανονικά τώρα προβλέπονται ε, εξηγήσει ψήφου, αλλά δεν έχει ζητήσει κανεί να κάνει επεξήγηση ψήφου, οπότε θα διακόψω τη συνεδρίαση μέχρι τι 3 και σα εύχομαι καλή σα όρεξη.